Allora diamo inizio ai nostri ξεκινήσουμε. Έχουμε τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών και ξεκινάμε λέγοντας ως συνήθως ότι η συνεδρίασή μας μαγνητοσκοπείται και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη σας δόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, άρα θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σας προτείνω μόνο να προσθέσουμε το εξής. Αύριο το πρωί θεωρήσα ότι οι ψηφοφορίες πρέπει να γίνουν στις 10.30 έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο από τις 9.30 στις 10.30 να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μάρτιν όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 90 του κανονισμού, καθώς επίσης και την έκθεση του κυρίου Γκουαλτιέρη όσον αφορά την τροποποίηση της οργανικής Συμφωνίας σχετικά με το Μητρό Διαφάνειας. Με την μικρή λοιπόν αυτή τροποποίηση που σας προτείνω και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Σας υπενθυμίζω ότι ο συνάδελφος Σέπφλιν διορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εισηγητής όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για την ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και ενστάσεις, επομένως συγκρίνεται και αυτός ο διορισμός. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η πρώτη ακρόαση Σύμφωνα με την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, όσον αφορά λοιπόν το δικαίωμα για το νερό, προβλέπεται για τις 17 Φεβρουαρίου 2014. Η δική μας η Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται άμεσα για το ζήτημα αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ έλαβα μια πρόσκληση για την ακρόαση αυτή από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και μπορείτε, μπορεί κάποιος εφόσον να το θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση. Πέρα από τον κύριο Χέφνερ που είχε την πρωτοβουλία για, την, το ζήτημα αυτό στο παρελθόν, οποιοδήποτε μπορεί στα πλαίσια του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει στην τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπεται από αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Λοιπόν, από τις 3 ως 6.30 το απόγευμα στις 17 Φεβρουαρίου 2014 και στην αίθουσα Γιάν 4Q2. Εγώ μάλιστα μάλλον θα συμμετάσχω. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά σας έχουν διανεμηθεί. Πρόκειται για τα πρακτικά της 25ης 26ης Νοεμβρίου 2013 και της 16ης 17ης Δεκεμβρίου 2013. Αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, τότε θεωρούμε ότι θα εγκριθούν και τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα εδώ είναι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εγώ είμαι ο εισηγητής για το ζήτημα αυτό. Θα θυμάστε ότι ήδη σας παρουσίασα τις βασικές ε, κατευθυντήρες γραμμές της έκθεσής μου στις 21 ε, Ιανουαρίου. Άκουσα μάλιστα και τις δικές σας παρατηρήσεις και ελπίζω ότι τις έχω συμπεριλάβει στο γραπτό κείμενο που έχετε μπροστά σας. Έγινε και συνεθρίαση της ΚΟΖΑΚ, όπως γνωρίζετε στην Αθήνα, την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρο πριν από δύο εβδομάδε και στη συνεδρία σε αυτή λοιπόν στην Αθήνα εγώ ήμουν εισηγητή ακριβώ για το ζήτημα αυτό. Σχέσει δηλαδή ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μου δόθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να ενημερώσω τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων για το ζήτημα αυτό. Η δική μου η έκθεση βέβαια είναι η πρώτη για το ζήτημα αυτό. Όπως ξέρετε έπρεπε να λάβω υπόψη μου και το έκανα αυτό ιδιαίτερα ευχάριστα, τις παραλυθούσες εκθέσεις που έχουμε για το ζήτημα αυτό από το 1997, από την έκθεση του 2002 και την έκθεση του 2009. Το 1997 είχαμε την έκθεση Nate Shooter Brock, αργότερα την έκθεση Ναπολιτάνο και αργότερα την έκθεση Brock το Μάιο του 2009. Έλαβα λοιπόν υπόψη μου όλες τις εκθέσεις αυτές και η δική μου η πρόθεση, την οποία έχω εκφράσει στο γραπτό αυτό κείμενο και μπορείτε προφανώς να υποβάλλετε και περαιτέρω τροπολογίες για να τη βελτιώσετε την έκθεση αυτή, η δική μου πρόθεση, επαναλαμβάνω, ήταν να ερμηνεύσω σαστικά την υφιστάμενη κατάσταση. Και ο στόχος μου ήταν να ερμηνεύσω λοιπόν τα όσα ήδη υφίστανται από θεσμικής πλευράς όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λέω σε κάποιο σημείο της εκθεσής μου ότι υπάρχει πραγματικά ένα κοινοβουλευτικό ευρωπαϊκό σύστημα και στο ευρωπαϊκό αυτό κοινοβουλευτικό σύστημα ανήκουν προφανώς και τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν πρέπει να αποτελούν ένα εξωτερικό στοιχείο του συστήματος αυτού, αλλά ένα αναπόσπαστο σύστημα, ένα αναπόσπαστο μέρος αυτού του συστήματος, όπως ακριβώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως είπα και στην προηγούμενη εισήγησή μου, βλέπουμε ότι η ίδια η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει μία ενεργό συμμετοχή, όχι μόνο απλώς έναν έλεγχο και έναν ρόλο επιτήρησης, αλλά μία ενεργό συμμετοχή στα ευρωπαϊκά ζητήματα από τα εθνικά κοινοβούλια. Και επίσης, τα εθνικά κοινοβούλια δεν προβλέπουν μόνο έναν έλεγχο όσον αφορά την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων των εθνικών θεσμικών οργάνων, αλλά συμβάλλουν σε ένα πραγματικό, επικοδομητικό, πολιτικό διάλογο και υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την ανάληψη δράσης. Επιβεβαιώνω λοιπόν στην έκθεσή μου ορισμένα πράγματα τα οποία εφίστανται ήδη. Επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία λέγονται και σε προηγούμενες εκθέσεις. Λέμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν πρέπει να αποτελούν μια τρίτη βουλή. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το έχουν πει και άλλοι οι ε, στο παρελθόν δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τρίτη βουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συστήματος, γιατί τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν τελικά στην δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος τους λοιπόν της δημοκρατικής αυτής νομιμοποίησης έχει να κάνει με την δεύτερη αν θέλετε βουλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι στο Συμβούλιο. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν ελέγχοντας τις ε, κρατικές κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις ουσιαστικά νομιμοποιούν δημοκρατικά το ρόλο του Συμβουλίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται τα εθνικά κοινοβούλια πριν και μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και πριν τα Συμβούλια των Υπουργών. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα επιπλέον καθήκον των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πέρα από το καθήκον αυτό όμως έχουμε και το καθήκον της ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία πρέπει να αποτελεί όχι συνεργασία μεταξύ δύο απομονωμένων οργάνων, αλλά μια επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα σε δύο απόσπαστα τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συστήματος. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, κατά τη δική μου την άποψη, διαδραματίζουν ένα ρόλο συμβουλευτικό, συμβάλλουν στην προκαταρκτική νομοθετική διαδικασία και ουσιαστικά εμπλουτίζουν με το έργο τους το έργο το οποίο κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πάντα παρόν στις συνεδριάσεις, στις διακοινοβουλευτικές που λαμβάνουν χώρα. Και έτσι λοιπόν και στις διάφορες διασκέψεις που βλέπουμε, όσον αφορά και παράδειγμα την ΚΟΣΑΚ ή και σε άλλες διακοινοβουλευτικές συνδιασκέψεις, όπως για παράδειγμα για την οικονομική διακυβέρνηση, για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας, βλέπουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συμμετέχει πάντα. Η συνεργασία αυτή στο ευρωπαϊκό αυτό κοινοβουλευτικό σύστημα θα πρέπει να εκφράζει με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο μια θετική άποψη όσον αφορά τις ε, νέες αυτές διακοινοβουλευτικές διασκέψεις που έχουν θεσπιστεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ρόλο καθοδήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις νέες αυτές διακοινοβουλευτικές διασκέψεις και λέγεται επίσης και στο κείμενό μου ότι θα πρέπει να συζητώνται πλέον κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στις διακοινοβουλευτικές αυτές συνεδριάσεις και λέμε επίσης ότι η ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται με ένα συγκεκριμένο όμως καθήκον πλέον, μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα η ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εννοώ είναι πώς προοδεύει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Να γίνεται αυτό ουσιαστικά σε μηνιαία βάση. Στην έκθεση αυτή γίνονται και κάποιες περαιτέρω προτάσεις πέρα από την απλή διαπίστωση των πραγμάτων ως έχουν. Λέμε επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την διακοινοβουλευτική συνεργασία. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να μπορούν να προετοιμάζουν τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και ένα ακόμα σημείο το οποίο θέτω με την έκθεση με αυτή είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου υπαριθμών 9, καθώς επίσης και το άρθρο 130 του κανονισμού μας, έτσι ώστε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να υπάρχει μια επίσημη διοργανική πλέον διακοινοβουλευτική συνεργασία, ε, συμφωνία με συγχωρείτε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κατά αυτόν τον τρόπο μέσω μιας ε, διακοινοβουλευτικής τέτοια συμφωνίας θα θεσπίζονται με τρόπο επίσημο οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και μεταξύ αυτών συνεργασία. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία της εκθεσής μου και προφανώς μπορείτε τώρα να πάρετε το λόγο για να κάνετε παρατηρήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω να καταγράψω και τις δικές σας προτάσεις και με αυτές να εμπλουτίσω στην εκθεσή μου. Επίσης, θα πρέπει οι προτάσει αυτές στη συνέχεια να εμπλουτίσουν ακόμα και τις συνεδριάσεις που γίνονται για την διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ντάφ έχει πρώτος το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για το σχέδιό του. το οποίο έλαβα πριν το μεσημεριανό και τώρα μόλις διάβασα. Περιέχει πολλά θέματα ουσίας. Και αξίζει να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το πώς θα το χειριστούμε στο Κοινοβούλιο. Σε προηγούμενη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό εξέφρασα τη σκέψη ότι ίσως είναι πολύ νωρίς μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για να σκεφτούμε μια αναθεώρηση των ρυθμίσεων που έχουμε θεσπίσει όσον αφορά τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι ακόμα προσπαθούμε να κατασταλάξουμε στο πείραμα αυτό, προσπαθώντας να βρούμε πράγματα που θα λειτουργήσουν καλά στην πράξη και καταργώντας πράγματα που δεν λειτουργούν. παρότι συχνά φαίνεται να είμαι από την πλευρά αυτών που θέλουν να επιταχύνουν όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά. Σίγουρα, προτού να αποφανθούμε πάνω στα θέματα αυτά και υπαγορεύσουμε οποιαδήποτε βελτίωση του πρωτογενούς ή δευτερογενούς δικαίου θα πρέπει να έχουμε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να ακούσουμε τις δικές τους εμπειρίες και νομίζω ότι θα λάβουμε πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Νομίζω ότι κάποια Εθνικά Κοινοβούλια έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην πρόκληση τη συνθήκης της Λισαβόνα και θέλω να αναφέρω το Bundestag ως παράδειγμα ενός τέτοιου κοινοβουλίου που έχει αγωνιστεί να βελτιώσει την επεξεργασία ευρωπαϊκών θεμάτων. Βρίσκουμε όμως και αρκετά εθνικά κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν, να αναπαθμίσουν τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά θέματα. Όλα όμως τα κοινοβούλια νομίζω θα πούν ότι αγωνίζονται για την συνεργασία μαζί μας, ότι αυτό απαιτεί πολλούς πόρους και χρόνο για να ανταποκριθούν σε αυτά που τους ζητάμε. Τα οποία είναι σημαντικά. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε εκπόνηση έκθεσης της ΑΦΚΟ πάνω στο θέμα αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε όλες οι άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Όλες οι επιτροπές έχουν τις δικές τους εμπειρίες όσον αφορά τη συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια και νομίζω ότι θα προκαλέσουμε αρνητική αντίδραση εάν προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση χωρίς να συμμετέχουν οι άλλες επιτροπές, ως άλλωστε σημαντικοί ενδιαφερόμενοι. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι γενική. Σε καμία ομοσπονδιακή δομή τα κοινοβούλια των επιμέρους κρατών δεν παίζουν ρόλο στην ομοσπονδιακή διακυβέρνηση. Η προσέγγιση που θεσπίζει η συνθήκη της Λισαβόνας και που ενθαρρύνει εδώ ο πρόεδρος μας είναι μια μορφή διακοινοβουλευτικής συνεργασίας που φέρνει τα εθνικά κοινοβούλια άμεσα μέσα στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, υπάρχει δηλαδή αυτή η λειτουργία ελέγχου και κάποια κοινοβούλια ξέρουμε ότι είναι δυσαρεστημένα που δεν μπορούν να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στην επί της εξέταση της ποιότητας των νομοθετημάτων. Είναι όμως γεγονός ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη διάκριση, από το διαχωρισμό των εξουσιών, ούτε να μπλέξουμε το ομοσπονδιακό με το εθνικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο. Θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και δεν θα ήταν πολύ εύκολο να εξηγηθεί στον ψηφοφόρο που θα πρέπει να βλέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις νομοθετικές εξουσίες του δικό μας Κοινοβουλίου και την νομιμοποίηση των, ε, δικό των δικών τους εθνικών κοινοβουλίων. με την πρώτη ματιά που έριξα στο κείμενο αυτό, διαπίστωσα ότι ο πρόεδρος λέει ότι δεν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο σώμα, ένα νέο φορέα, ένα νέο θεσμικό όργανο. Προτείνει η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων να επισημοποιηθεί, πράγμα που ακριβώς αντιφάσκει με αυτό που είπε. Και ανησυχώ ότι αυτή η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων ε, θα ξεφύγει από αυτό που είναι προς το παρόν και θα γίνει κάτι άλλο. Οι θέσεις των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Ο ρόλος τους, ε, συγγνώμη, διαφέρει πολύ. Είναι μερικοί που απλά παίζουν έναν τυπικό ρόλο Προέδρου. Ενώ άλλοι κατέχουν πολλές εξουσίες όσον αφορά τη διαμόρφωση του θεματολογίου και της πολιτικής του Κοινοβουλίου τους. Είμαι λοιπόν πολύ επιφυλακτικός σε όλα αυτά. Λέτε επίσης κύριε Πρόεδρε, ότι η ΚΟΣΑΚ θα πρέπει να αναλάβει πιο εξειδικευμένο ρόλο, να αποτελεί φόρουμ για συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτός ο ρόλος είναι πολύ γενικός. Και αν απαιτείται απλά συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ευρώπης, θα υπάρξει σημαντικός βαθμός δυσαρέσκειας. Και η συζήτηση αυτή θα απέχει πολύ από τις πρακτικές και νομοθετικές εργασίες της Ένωσης. Αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να βρούμε μια σοβαρή λειτουργία, ε, έναν σοβαρό ρόλο για την ΚΟΖΑΚ. παρουσιάζεται την ιδέα ενός επίσημου μέσου που να συνυπογράφεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από μας. Αυτή είναι μια καινοτόμα ιδέα που θα απαιτήσει πολύ προσεκτική σύνταξη και αιτιολόγηση. Το ένστικτό μου μου λέει ότι αν το εξετάσουμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι κάτι που δεν θα λειτουργήσει. Διότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να εξουσιοδοτήσουν εκπροσώπους να λαμβάνουν αποφάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ευρωπαϊκή διάσταση δηλαδή. Κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο οποιαδήποτε δέσμευση με επίσημη συμφωνία με άλλα κοινοβούλια, πόσο μάλλον με εμάς πέρα από τα πλαίσια της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, είναι πολύ μεγάλο βήμα. Κάποια κοινοβούλια θα το κάνουν αυτό πολύ πιο ευχαρίστως από άλλα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι το κοινοβούλιο του Westminster, το οποίο γνωρίζω αρκετά καλά, θα τρομάξει με την ιδέα να δεσμευτεί με μια πολυμερή διακοινοβουλευτική συμφωνία. Και μια τελευταία παρατήρηση. εάν είναι να μιλάμε για το, εθνικό, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και την ε, κοινή εξωτερική και πολιτική και πολιτική άμυνας και τη συνεργασία στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε την πολυεπίπεδη δομή των θεμάτων αυτών. δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια σε, όλους τους, ε, σε όλες τις βαθμίδες συνεργασίας. Υπάρχουν δηλαδή περιφερειακές ομάδες. Αυτό το γεγονός λοιπόν θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ρυθμίσεων για την διακοιλοβουλευτική συνεργασία. Λυπάμαι που είμαι επικριτικός, αλλά φοβάμαι λίγο με το φάκελο αυτό. Θα ήθελα όμως να επενέσω τον Πρόεδρο για την τολμηρή πρωτοβουλία του. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, uh, uh, Ο Ρίκο Γερέρο, που είναι μόνιμο μέλος της ε, Επιτροπής, μου ζήτησε να σας ενημερώσω για την άποψή του. Το βασικό σημείο της έκθεσης είναι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εθνικά κοινοβούλια ανήκουν στο εθνικό πολιτικό σύστημα της κάθε χώρας, αλλά και ταυτόχρονα στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Τουλάχιστον από την Συνδίκη Λισαβόνας και μετά. Σήμερα αυτό ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο από νομικής πλευράς αλλά και από πολιτικής πλευράς. Ξεκινώντας από τη δεύτερη, την πολιτική πτυχή, η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορεί να ενθαρρύνει περαιτέρω ολοκλήρωσή τους στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα και θα μπορούσε επίσης να συνεισφέρει και στην βελτίωση της ε, νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι, στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό την εποχή της κρίσης που ζούμε και εν ώψη των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών. Από νομικής πλευράς, από την άλλη μεριά, το άρθρο 12 της Συνδική Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλου 1 και το πρωτόκολλο 1 αναγνωρίζουν το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν θεσμοθετούν το ρόλο αυτό με την έννοια ότι ε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως, ε, ε, με, με, την έννοια ότι ούτε αποτελούν τρίτο πόλο, ούτε αποτελούν ένα ανεξάρτητο όργανο στο, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γι' αυτό το λόγο τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συνεργάζονται με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να αντιμάχονται, να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ή να αλληλοπικαλύπτονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άλλη μεριά δεν δίνει λογαριασμό στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, αντιθέτως, ε, ε, ε, είναι υπεύθυνο εναντί των Ευρωπαίων πολιτών. Τα Εθνικά Κοινοβούλια από την άλλη μεριά είναι υπεύθυνα, μάλλον συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τα θέματα τα οποία αποτελούν αρμοδιότητά του σύμφωνα με τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Εθνικά Κοινοβούλια όμως ε, δίνουν νομική βάση και νομιμοποίηση το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική. Ενώ επίσης υφίστανται διάφορες διατάξεις στην συνθήκη που προβλέπουν την συμμετοχή των Αθηνικών Κοινοβουλίων όπως για παράδειγμα ε, στην, ε, ε, αποδίδεται στα κράτη, στα εθνικά κοινοβούλια ο ρόλος της συνένεσης προκειμένου ορισμένε αποφάσεις της Ευρωεξένωσης να μπορούν να εφαρμοστούν. Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου 1 και το άρθρο 130 της συνθήκης προβλέπουν μια διοργανική συμφωνία έτσι ώστε να θεσμοθετηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, θα πρέπει να γίνει ε, να δοθεί ένας καινούριο ορισμός στην αποστολή της ΚΟΖΑΚ. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαρθρωμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ΚΟΖΑΚ ενώ οι διασκέψεις θα πρέπει να οργανώνονται, να υλοποιούνται για συγκεκριμένα θέματα, εξωτερική πολιτική, Eurojust και Europol, οικονομική διακυβέρνηση κλπ όχι ε, επιγενικών ε, ε, θεμάτων ούτε για γενική συζήτηση. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ο προσανατολισμός και διάρθρωση στην διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου ο ρόλος τους να είναι σαφής, καθαρός και να αποφεύγουμε παρεξηγήσεις, ανταγωνισμούς αντιζηλίες κλπ. Από νομικής και πολιτικής πλευράς λοιπόν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Η έκθεση λέει θα γίνει στην επόμενη θητεία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή μας στην ε, επόμενη κοινοβουλευτική μας θητεία. Το σχέδιο έκθεση είναι μια καλή βάση για την ανάλυση του ζητήματος συμφωνούμε ιδιαίτερως με, με την ιστορική εξέλιξη της ε, συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την εμπειρία των Εθνικών Κοινοβουλίων για το σύστημα ε, έγκαιρης ειδοποίησης, σε ό,τι αφορά την αρχή της επικορικότητας, για την συμμετοχή των Εθνικών κοινωνιών σε ορισμένα θέματα ευρωπαϊκή δραστηριότητα, όπω για Eurojust, Europol, Αλία, ε, συγγνώμη, εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλεια, οικονομική διακυβέρνηση κλπ. Ε, επίσης, η COSAC θα πρέπει να ασχολείται με συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων και όχι σε γενική συζήτηση όπω γίνεται μέχρι τώρα. Πιστεύουμε όμω ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν και ορισμένα ζητήματα στην έκθεση ή να αναλυθούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, οι διακυβερνητικές διασκέψεις που δίνουν φωνή στα εθνικά κοινοβούλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση να αναλυθουν περαιτερω για παραδειγμα οι διακυβερνητικέ διασκεψεις που δινουν φωνη στα εθνικα κοινοβουλια σε ευρωπαικο επιπεδο η προταση να παμε πιο μακριά και να θεσμοθετήσουμε αυτές τις σχέσεις δεν θα πρέπει να καταλήξει στην δημιουργία ενός μηχανισμού διακοινοβουλευτικής λήψης αποφάσεων. Δεύτερον, καλωσορίζουμε την ιδέα του νησιγητή περί της δημιουργίας της υπογραφής μιας ε, συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων προκειμένου να διαρθρωθεί καλύτερα η συνεργασία, ανταλλαγή ε, πληροφοριών κλπ. Παρ' όλα αυτά και πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι δημιουργείται μια καινούργια ενδιάμεση δομή, ένα καινούργιο ενδιάμεσο επίπεδο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ανάμεσα μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, τα, και την εθνική πολιτική σκηνή. Η βελτιωμένη συνεργασία, προκειμένου να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ε, εθνικών κοινοβουλίων, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Τέλος, το σημείο 3 της έκθεσης αναφέρεται σε πρακτικές προτάσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό το τμήμα θα μπορούσε να ε, ενισχυθεί με πρόσθετες ιδέες και πρακτικές προτάσεις και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί ταυτόχρονα όμως και πιο ρεαλιστικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μορέιρα. Ο κύριος Σέπφλιν έχει τώρα το λόγο. Thank you, Chair, and indeed, thank Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα ήθελα να θέσω μια σειρά ερωτήσεων. Δεν διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση, την έλαβα μόλις πριν το μεσημεριανό γεύμα, αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Το η έκθεση μιλάει για ένα ευρωπαϊκό κοινοπλευτικό σύστημα. Πρόκειται όμως πραγματικά για σύστημα. Μήπως στην πραγματικότητα είναι μία άνηση πολυεπίπεδη σχέση, μία σειρά ασυμμετριών. Στην περίπτωση αυτή δεν νομίζω ότι η λέξη σύστημα είναι ιδιαίτερα πιστική. Δεύτερον, η έκθεση μιλάει για έναν μόνιμο διάλογο. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για διάλογο. Συμμετέχουν πολύ περισσότεροι από δύο ε, συμμετέχοντες. Ε, υπάρχει η λέξη πολύ λόγος, αλλά το θέμα είναι ότι είναι μια συζήτηση σε πολλά επίπεδα και Επίσης, πόσο αποτελεσματικός είναι αυτός ο διάλογος στην πραγματικότητα. Τα εθνικά κοινοβούλια πώς βλέπουν το ρόλο τους στο συγκεκριμένο σύστημα. Έχει εξερευνηθεί αυτό. Και σε συνέχεια, και εδώ φτάνουμε στον πυρήνα της έκθεσης, πώς θα πρέπει να, κατανοήσουμε την, ε, τον διαχωρισμό, την σχέση κυριαρχίας ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση για το εγγύς μέλλον. Και αυτή η δομή είναι σταθερή, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ε, μεταβάλλεται μία προς τη μία κατεύθυνση, μία προς την άλλη. Ε, όχι τόσο πολύ με νομικούς όρους, αλλά πολιτικούς όρους. Και σε προηγούμενες συναντήσεις έχουμε μιλήσει για τις ε, διάφορες ε, δυνάμεις. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επανέλθει η κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο, άλλοι που θέλουν να την φέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι εξορισμού πιο διαρρεμένα από ότι είναι η, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασχολούνται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά. Τα εθνικά κοινοβούλια όμως ε, νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν την καθημερινή ζωή και τους διάφορους συνασπισμούς που υπάρχουν σε κάθε πολιτικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι αυτές οι δύο πλευρές μπορούν να συμφιλειωθούν. Νομίζω ότι και αυτό αποτελεί ένα μέρος της ασυμμετρίας στην οποία αναφέρθηκα. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι τι γίνεται με τα περιφερειακά κοινοβούλια πώς ε, ταιριάζουν αυτά στο σύστημα αυτό. Και τέλος, μια σκέψη. Ίσως θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό ανάλογα με το αν μπορούμε να μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πολιτεία, μια ευρωπαϊκή πολιτική οντότητα. Ο κύριος Νταφ μίλησε για ε, ομοσπονδία. Δεν νομίζω ότι ο όρος του φεντεραλισμού ταιριάζει εδώ, διότι αυτό που έχουμε εδώ είναι τόσο ρευστό. Δεν είναι ούτε ομοσπονδία ούτε συνομοσπονδία. Τι ακριβώς είναι. Και κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ε, αυτό αποτελεί, αυτά τα ερωτήματα αποτελούν μέρος της εκθέσης σας, κύριε Πρόεδρε. Parola adesso al Messerschmidt Thank you, Chair. I will not... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρότι μπαίνω σε πειρασμό, δεν ε, θα αναφερθώ στην Ομοσπονδία ή στην Ομοσπονδία, θα περιοριστώ στην έκθεση. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα και σημαντικά θέματα, τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Ένα από αυτά είναι φυσικά ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων σύμφωνα με τη συνθήκη. Αναφέρεται η αρχή της επικουρικότητας και η λειτουργία ελέγχου. Ωστόσο, έχει προκύψει ένα πρακτικό πρόβλημα στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ένα καθαρά οργανωτικό θέμα. Οι 8 εβδομάδε που έχουν στη διάθεσή του, που νομίζω ότι είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για πολλά κοινοβούλια, πόσο μάλλον που έχουν και άλλε δουλειέ. Αυτό συχνά αναφέρεται στην ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό λοιπόν και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν θυμάμαι τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορέσουν να οριστικοποιήσουν ε, κάποιο νομοθέτημα σε 8 εβδομάδες. Δεν ε, θα έβλεπε λοιπόν αν τα εθνικά κοινοβούλια είχαν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μια βασική αρχή της νομιμότητας. Εάν δεν γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας στην νομοθεσία, είναι κατά της συνθήκης να συνεχίσουμε ε, στην ε, υιοθέτηση της ε, νομοθεσίας αυτής. Οχτώ εβδομάδες λοιπόν δεν αρκούν. Δεύτερον, η ΚΟΣΑΚ. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Ντάφε και άλλοι ομιλητές σχετικά με το ρόλο της ΚΟΣΑΚ. Αμφιβάλλω εάν εναπόκειται σε εμά να εκπονήσουμε έναν ορισμό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα μεταξύ των 29 κοινοβουλίων της ΚΟΣΑΚ. Είμαστε απλά ένα κοινοβούλιο μεταξύ των άλλων. Ε, έτσι έχει αποφασιστεί. Γιατί λοιπόν να ορίσουμε εμεί τι θα είναι η ΚΟΣΑΚ, μήπω θα ήταν πιο φρόνιμο να ανοίξουμε μια συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να έχουμε νέο ορισμό, να καθορίσουμε εκ νέου τις, ε, τα θέματα που ενδιαφέρουν την ΚΟΣΑΚ. Συμφωνώ ότι σήμερα όλα είναι πολύ θολός και ασαφής ο ρόλος της ΚΟΣΑΚ και αυτό είναι κρίμα. Εγώ θα προτιμούσα να έχω ένα θεσμοποιημένο σώμα, ωστόσο καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά ας έχουμε τουλάχιστον ένα επίσημο φόρουμ όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συναντηθεί με τα άλλα εθνικά κοινοβούλια και να συζητάει θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παρότι, κύριε Πρόεδρε, Πιστεύω ότι είναι πολύ περιορισμένο να ζητάμε από την ΚΟΣΑΚ να ασχολείται μόνο με την κατάσταση της Ένωσης. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτό συνδέεται με την ομιλία του ε, Πρόεδρου της Επιτροπής, ε, την ομιλία State of the Union για την κατάσταση της Ένωσης. Υπάρχουν όμως πολλά τεχνικά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στην νομοθετική διαδικασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτή ήταν η δεύτερη παρατήρηση. Και η τρίτη παρατήρηση, πολύ σύντομα, έχει να κάνει με την IPEX, ε, την οποία συμβουλεύομαι ε, όχι πολύ συχνά για να δω τι γίνεται με τις ε, διαδικασίες ελέγχου στα Εθνικά Κοινοβούλια και μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργάζεται κανεί με το εργαλείο αυτό. Πολύ συχνά δεν έχουμε μετάφραση των εκθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να διαβάζω βουλγάρικα και κυπριακά. Δεν μπορώ ε, λοιπόν να αποφασίσω αν συμφωνώ με τα κοινοβούλια αυτά, τα οποία σύμφωνα με τη συνθήκη έχουν ε, ε, εξουσίες, έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν χειριζόμαστε σωστά την αρχή της επικουρικότητας ή όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν οικονομικού και άλλου πόρου για την ΑΕΠΕΞ. σω αυτό προσπαθείτε να μα πείτε στο σημείο 27, όπου λέτε ότι πρέπει να έχουμε ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού. Εάν ναι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει τονιστεί, ώστε να λειτουργεί καλύτερα αυτή η ιστοσελίδα στο μέλλον. Για, εάν θέλουμε δηλαδή να σεβαστούμε την αρχή αυτή και να πάρουμε στο σοβαρά τη συνθήκη. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει που είχα προ εσά, κύριε Πρόεδρε ως εισηγητή τη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπρόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η έκθεση κατά βάση ε, θέτει το ερώτημα ποιο είναι ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η ερώτηση δεν είναι τόσο χαζή όσο φαίνεται, δεδομένη τη μεταφορά των νομοθετικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βέβαια, ε, στην περίπτωση των οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να μεταγράψουν τι οδηγίε αυτέ. Όμω είναι προφανέ ότι οι αποκλειστικέ αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβούλιων συρρυκνώνονται και θα συνεχίσουν να συρρυκνώνονται γνωρίζουμε πλέον ότι το βασικό καθήκον των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι να ελέγχουν την κυβέρνησή τους που αντιπροσωπεύει τη χώρα στο Συμβούλιο. Ε, τα Εθνικά Κοινοβουλία θα έπρεπε λογικά να είναι υπεύθυνα και να δοτούν έναντι του, του εκλογικού του σώματος και να παίρνουν εντολές από αυτό. Όμως στην πραγματικότητα φαίνεται ότι ο ρόλος του πλέον είναι να ελέγχουν το Συμβούλιο και να αποφεύγουν τα, ε, η κυβέρνησή τους να ε, παίρνει θέσεις οι οποίες είναι παράλογες. Ε, τώρα, αν κατάλαβα καλά, ο κ. Νταφ είπε ότι τα κράτη μέσα σε μια ομοσπονδία δεν έχουν ρόλο να παίξουν σε ομοσπονδιακά θέματα. Είναι ανοιχτό ε, φίλο τη ομοσπονδιακή Ευρώπη. Όμω, όχι, δεν είμαστε όλοι μα ε, μάλλον ε, πολλοί άλλοι δεν είναι τόσο ανοιχτοί και τόσο ειλικρινείς. Ε, έγινε προσπάθεια η λέξη ομόσπονδος ή ομοσπονδιακός να συμπεριληφθεί στην συνθήκη του Μάστρικτ που στην πραγματικότητα έγινε και συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. βέβαια, ο Τζον Μέιτζορ επέμεινε να μην συμβεί αυτό και δεν συνέβη, ε, διαγράφηκε η λέξη αυτή. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Ε, η άποψή μου είναι όμως ότι η, τα κράτη θα πρέπει να επιστρέψουν στην πηγή και να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των δικών τους λαών και όχι μιας ε, ομοσπονδιακής Ευρώπης. Τα εθνικά κοινοβούλια παίρνουν εντολή από τον λαό για μια όλο και πιο διευρυμένη ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λέει η έκθεση. Όμως ε, ε, υπάρχει το κίνδυνος να παραπλανηθούν από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι λένε, σχεδόν ότι τα εκπροσωπούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην θυμώσετε, εάν πριν περάσω στο περιεχόμενο, αναφέρω ότι έχουμε εδώ μια έκθεση με ένα πάρα πολύ σημαντικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στην ε, Επιτροπή, αλλά έχουμε λάβει το κείμενο λίγες ώρες πριν. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να συζητήσει κανείς γι' αυτό και θα είμαι σύντομος. Η έκθεση είναι σύντομη, τη λάβαμε όμως ε, τελευταία στιγμή και λυπάμαι γι' αυτό, διότι ειδικά το θέμα αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό κάποιες σύντομες παρατηρήσεις από τη δική μου πλευρά. Πιστεύω ότι είναι καλό και χρήσιμο ότι εξηγείται η νομική βάση στη συνθήκη ότι εξετάζει τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο σκεπτικός είμαι απέναντι στην πρόταση να έχουμε μια διοργανική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 28 διαφορετικούς παράγοντες δηλαδή. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας να βρούμε κατάλληλους τρόπους και να τους υιοθετήσουμε και γι' αυτό Λυπάμαι που δεν διατυπώνεται σαφέστερα η πρόταση εδώ. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στις προτάσεις σχετικά με τις διακοινοβουλευτικές συσκέψεις, διασκέψεις, όπου αναφέρεται όπου, ότι θα πρέπει να βελτιωθούν, όχι όμως το πώς. Εγώ συμμετείχα σε μια τέτοια διακοινοβουλευτική διάσκεψη και από μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων άκουσα να εκφράζεται αρκετή δυσαρέσκεια που συναντιόνται επί δύο-τρεις μέρες αλλά δεν έχουν την εντύπωση ότι μπορούν επί της ουσίας να συνεισφέρουν κάτι. Πιστεύω λοιπόν ότι με πιο σοφό, με πιο ικανό χειρισμό θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία και στο πλαίσιο αυτό μου φαίνεται καλό να ακούσουμε προτάσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, επί της μεθοδολογίας. Πώς δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μια τέτοια συνάντηση. Επικροτώ την πρόταση στο περιθώριο τέτοιων εκδηλώσεων να προβλέπεται οι πολιτικές ομάδες, τα πολιτικά κόμματα να συναντώνται ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και να μπορούν να παίξουν πιο ισχυρό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να δω προτάσεις σχετικά με την συνέχιση των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων στο, στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν υπάρχουν ε, μέχρι τώρα σαφείς κανόνες για κάτι τέτοιο και είναι σημαντικό στις συζητήσεις της Επιτροπής μας ε, να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τον ρόλο αυτών των διασκέψεων και να τον περιγράψουμε με περισσότερη ακρίβεια. Αυτά προς το παρόν. Πολύ σύντομα μόνο μπόρεσα να διαβάσω την έκθεση αυτή, διότι την έλαβα τελευταία στιγμή. Γι' αυτό επιφυλάσσομαι στο μέλλον να υποβάλω περισσότερες παρατηρήσεις, ενδεχομένως υπό τη μορφή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας καταρχάς. Σαφώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή τροποποίησης του κειμένου μέσω των τροπολογιών σας. Ο κύριος Χέφνερ είπε ότι λάβατε τελευταία στιγμή την έκθεση αυτή, αλλά έχει να κάνει και με την απόφαση που είχαν πάρει οι συντονιστές στο παρελθόν όσον αφορά την σύνταξη της έκθεσης αυτής διορίστηκε ο εισογητής, θυμάστε, με έναν τρόπο αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο. Έπρεπε να περιμένουμε να υποβληθούν πολλές διαφορετικές εκθέσεις και χρειάστηκε πραγματικά να κάνω τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρω πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή, αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι ε, ασχολήθηκα με ζητήματα τα οποία είχαμε αναλύσει καθόλου τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ήδη από το Βίλνιους και μετά, άμεσα ή έμεσα, συμμετέχοντας στην ΚΟΖΑΚ, έχω αναλύσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, κάποιους βασικούς αδρούς προσανατολισμούς αν θέλετε. Προφανώς πάντως υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης και τροποποίησης στις ιδέες αυτές. Θεωρώ κάποια πράγματα πάντως δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να τεθούν συζήτηση. Η γενικότερη αίσθηση που έχω εγώ από την κοινοβουλευτική μας αυτή θητεία όσον αφορά τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τόσο στην ΚΟΖΑΚ όσο και στην ομάδα εργασίας την οποία έχουμε για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και στα πλαίσια τη οποία είχα αποβάλει μια έκθεση, η γενικότερη αίσθηση που έχω είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια εν γέννη θέλουν να συμβάλλουν περισσότερο. Θέλουν ο λόγο του να μετράει περισσότερο. Μπορεί να υπάρχουν όντω ορισμένα κοινοβούλια τα οποία να έχουν ταχθεί κατά μια τέτοιας έντονη, αν θέλετε, προσχώρησή του στο ευρωπαϊκό σύστημα. Από την άλλη, υπάρχουν άλλα κοινοβούλια τα οποία έχουν ταχθεί σαφώ υπέρ μια τέτοια κοινοβουλευτική ολοκλήρωση. Εγώ ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσω απλώ μια αντιπροσωπευτική εικόνα των ε, πραγμάτων ω έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω κάποιε μεγαλεπίβολε προτάσει αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να καταλάβω κάπω πώ έχουν τα πράγματα και κάπω να τα οργανώσω, να του δώσω μια κάποια κατεύθυνση, έναν κάποιο προσανατολισμό. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου σε αυτή την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά το αίτημα των εθνικών κοινοβουλίων να μετράνε περισσότερο, πρέπει να δοθεί ως προς αυτό το αίτημα λοιπόν μία συγκεκριμένη απάντηση στα πλαίσια των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπερβούμε τα όσα λέγονται στη συνθήκη. Προφανώς είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα πρέπει να θεωρούνται σε καμία περίπτωση μια τρίτη βουλή, αφού το είπατε κι εσείς ε, οι ίδιοι, το έχετε γράψει και στο παρελθόν σε παρατηρήσεις που έχετε κάνει σε προηγούμενες εκθέσεις και προφανώς μπορείτε να το υποβάλλετε την ιδέα αυτή εκ νέου μέσω τροπολογιών. Νομίζω ότι ω προς αυτό συμφωνούμε. Εγώ ουσιαστικά προσπάθησα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ονομάζω στην εκθεσή μου Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα, που νομίζω ότι όντως υφίσταται κατά κάποιο τρόπο. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων δεν είναι, δεν ομοιάζουν με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων και άλλων κοινοβουλίων τρίτων χωρών. Φανταστείτε για παράδειγμα την συνέλευση ΑΚΕ ή άλλες μορφές κοινοβουλευτικής συνεργασίας που έχουμε. Τα κοινοβούλια αυτά δεν συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν σε αυτό το οποίο ονομάζω εγώ Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα. Επομένως συμμετέχουν πολύ πιο άμεσα και στον έλεγχο των Εθνικών Κοινοβουλίων προφανώς που είναι η βασική τους αρμοδιότητα, αλλά και στον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό ακριβώς θέλω να ευανθύνω. Αυτός ο πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να είναι ένας διάλογος ο οποίος να επηρεάζει τι αρμοδιότητε λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι τα εθνικά κοινοβούλια ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο μέσω του διαλόγου αυτού στη λήψη αποφάσεων που προφανώ θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς λέω ότι θεωρώ, θα, θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε πιο θετικά τα εθνικά κοινοβούλια, ότι δεν τροχοπεδούν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά τις εμπλουτίζουν με νέες ιδέες, με νέες προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, να καταφέρνουμε εγκαίρως να λαμβάνουμε τις ε, αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν προφανώς περισσότερο, αλλά πάντα στα πλαίσια αυτού του πολιτικού διαλόγου. Σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι θα πρέπει να υπερβούν τις αρμοδιότητες λήψη αποφάσεων που έχουν αυτή τη στιγμή και να μπουν στον τομέα, αν θέλετε, στα χωράφια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά μια άλλη παρατήρηση που ακούστηκε, πρέπει να σας πω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή ως έχει αποτελεί ένα απλό στάδιο προς μία όλο και πιο στενότερη ένωση. Αυτή, αυτός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ως προς αυτό πρέπει να συμβάλλουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν προφανώς κάποια εθνικά κοινοβούλια τα οποία μπορούν να αποφασίσουν να περιορίσουν τη διαδικασία αυτή, να παρεμποδίσουν τη διαδικασία αυτή. Είναι το απόλυτο δικαίωμά του. Σε καμία περίπτωση πάντω, Στη συνθήκη δεν λέγεται κάτι τέτοιο. Στη συνθήκη λέγεται ότι ο βασικό μα στόχο, πείτε το αυτό Ομοσπονδία, δεν ξέρω πώ θα το πείτε, ο γενικό μα στόχο είναι να προσπαθούμε να κινούμαστε προ μια πιο στενή ένωση. Προσπαθούσα λοιπόν μέσω της έκθεσης αυτής με τρόπο ιδιαίτερα ταπεινό ακριβώς αυτό να παρουσιάσω ως βασικό στόχο και να δώσω μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Θα ήθελα να αναφερθώ επίση στι παρατηρήσεις του κυρίου Ντάφα. Προφανώς, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποκρισταλωθεί τα πράγματα και δεν ξέρουμε ακριβώ ποια κατεύθυνση ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τα εθνικά κοινοβούλια. Και ουσιαστικά αυτό ακριβώς έγινε στα πλαίσια της Κόζακ τα τελευταία πέντε χρόνια. Και χαίρομαι που στα πλαίσια της ε, διάσκεψης των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων αποφασίστηκε να συζητηθεί και αυτή μας ακριβώς η έκθεση που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στην τελευταία κόζακ της Αθήνας ακριβώς αυτό το ζήτημα συζητήσαμε και κατά αυτόν τον τρόπο όλες οι επιτροπές ευρωπαϊκών θεμάτων των Εθνικών Κοινοβουλίων κατάφεραν να τοποθετηθούν για το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, όπως το κύριο Σταφ, σαφώς είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και προφανώς θα πρέπει να μπλακούν και οι υπόλοιπε επιτροπές. Κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της νομοθετικής αυτής θητείας να τοποθετηθούμε. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχαίουμε τις διάφορες αρμοδιότητες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχαίουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή και τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως το να χρησιμοποιούν τις πορτοκαλί-κίτρινες κάρτες, το να σταματούν πολλές φορές την όλη νομοθετική διαδικασία όταν θεωρούν ότι δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Μπορούμε να αναλύουμε κατά αυτόν τον τρόπο την κατάσταση χωρίς προφανώς να τροποποιούμε ή να θεωρούμε ότι απειλείται η συνθήκη της Λισαβόνας. Αναφέρθηκα στις ε, διακοινοβουλευτικές ε, διασκέψεις για την οικονομική, δια... στην οικονομική διακυβέρνηση ακριβώς επειδή σχετική απόφαση είχε ληφθεί και στην Βαρσοβία. Νομίζω ότι είναι θετική η πρόταση αυτή. Τώρα αν θέλετε εσείς να υποβάλλετε κάποια τροπολογία κατά μπορείτε να το κάνετε. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ε, πρότασης αυτής για μια διακοινοβουλευτική διοργανική συμφωνία. Κάποιοι τάχθηκαν υπέρ, άλλοι πάλι κατά. Εγώ δεν αναφερόμουν σε μια συμφωνία που θα προβλέπει νέες αρμοδιότητες. Δεν είναι δυνατό άλλωστε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεται μια νέα συνθήκη, τροποποίηση τη συνθήκης για να γίνει κάτι τέτοιο. Αναφερόμουν σε μια διοργανική συμφωνία διαδικαστικής φύσης όχι θεσμικής, ουσιαστικής φύσης. Να λέμε δηλαδή πότε, γιατί, κατά ποιο τρόπο θα διεξάγονται αυτές οι διακοινοβουλευτικές διασκέψεις που πολλές φορές συμβαίνουν και διοργανώνονται κάπως τυχαία. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες προκειμένου να διοργανώνονται καλύτερα και πιο συντονισμένα αυτές οι διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν θετικό το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί και με αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι έχω απαντήσει σχεδόν σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Σαφώς δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρανοήσεις, σαφώς δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Μορέιρα, αυτό όμως λέω και εγώ στις απόψεις που εκφράζω στην έκθεση. Προφανώς υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Να καταφέρουμε να δυναμώσουμε κάποιες προτάσεις. Εγώ προσπάθησα να είμαι κάπως ε, προσεκτικός. Ξέρω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ δύσκολο και ενδεχομένω το τμήμα αυτό των προτάσεων είναι και το πιο αδύναμο της εκθεσής μου. Θεώρησα και το παραλαμβάνω αυτό ότι βασικός στόχος της εκθεσής μου είναι να δώσω μια εικόνα, μια φωτογραφία αν θέλετε, της κατάστασης. Ξέρετε ότι αυτή η διοργανική συμφωνία ουσιαστικά προβλέπεται αυτή τη στιγμή και από τη συνθήκη. Αν δεν συμφωνούμε, ας τροποποιήσουμε και τη συνθήκη. Σε μια μελλοντική συνέλευση θα πρέπει να λέμε ότι θα αλλάξει το άρθρο 9 του πρωτόκολλου παριθμών 1. Κύριε Σέπφλιν, Σε ένα σημείο της έκθεσης λέμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα περιφερειακά κοινοβούλια και τα λοιπά. Και το έθεσα αυτό επειδή ακριβώ η παρατήρηση αυτή είχε γίνει και κατά τη συζήτηση προηγούμενων εκθέσεων. Δεν ξέρω βέβαια πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τα περιφερειακά κοινοβούλια. Συμφωνώ όμως μαζί σας, ας προσπαθήσουμε από κοινού να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το ρόλο τους πιο επικοδομητικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπατε εσεί στη συνέχεια, κύριε Μπρόνς, αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία ομοσπονδιακή ή μη κατεύθυνση. Μα αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται και το οποίο τίθεται και στι επόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ. Για ποιο λόγο να μην το θέσουμε και εμεί στα πλαίσια τη έκθεση αυτή. Εν τέλει, κύριε Μέσσερμιτ, οι οκτώ αυτέ εβδομάδε, σύντομο χρονικό διάστημα, όντω συμφωνώ, το έχουν πει και πολλοί άλλοι. Μπορείτε λοιπόν να υποβάλλετε μια τροπολογία προκειμένου να επιμηκυνθεί η περίοδος αυτή. Εγώ θεωρώ θα μπορούσε να γίνει αποδεχθή μια τέτοια τροπολογία. Σας ευχαριστώ επίσης ε, γιατί συμφωνείτε με το να θεσπιστεί μια νέα γραμμή του προπολογισμού. Είπα ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο την πλατφόρμα IPEX. Συμφωνώ μαζί σα, Και ένα λεπτό τώρα ζήτημα. το ζήτημα των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων και πώς θα μπορούσαν να διαρθρωθούν. Δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει απλώς να συμμετέχει ως ένα απλό τμήμα των διασκέψεων αυτών. Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους Ευρωπαίους πολίτες κατά τρόπο άμεσο και καθολικό. Πρέπει λοιπόν να προωθεί αυτό πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η παρουσία λοιπόν των άλλων εθνικών κοινοβουλίων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως παρουσία συνομοθετών. Ουσιαστικά οι κοινοβουλευτικέ αυτέ διασκέψει δεν έχουν ως στόχο να αποδυναμώσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακριβώ το αντίθετο, να ενισχύσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως στόχο αυτέ οι διακοινοβουλευτικέ διασκέψει. Να τον ισχύσουν τι στιγμέ εκείνε που πρέπει να κάνει κάποιε επιλογέ, να πάρει συγκεκριμένε νομοθετικέ αποφάσει είναι πολύ σημαντικό να μπορούν στη δικασία αυτή να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια, και αυτό λέγεται γενικότερα στην έκθεση, ανέκαθεν εκπροσωπούσαν μια ευρωπαϊκή συνείδηση και θα πρέπει να εκπροσωπούν αυτή την ευρωπαϊκή συνείδηση. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη-μέλη και σε κάποια εθνικά κοινοβούλια η ευρωπαϊκή αυτή συνειδητοποίηση δεν είναι τόσο έντονη όσο σε κάποια άλλα. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θεωρώ πάντως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να τονίζεται από τη νέα δομή που θα δοθεί στις διακοινοβουλευτικές αυτές, αυτές διασκέψεις ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να απαντήσω τέλος στον κύριο Χέφνερ. Όσον αφορά την καθυστέρηση στην υποβολή της έκθεσης αυτής, έδωσε μια κάποια αιτιολόγηση όσον αφορά την αγανάκτηση των συναδέλφων από τα εθνικά κοινοβούλια που θεωρούν ότι ο λόγος τους δεν ακούγεται, η φωνή τους δεν ακούγεται αρκετά. Μα συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό σύστημα στο οποίο να συμμετέχουν δυναμικά και τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι τόνισα κατά τρόπο θετικό τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμπλέξουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τώρα, Είπατε ότι ενδεχομένως η συμμετοχή των 28 διαφορετικών εθνικών κοινοβουλίων να περιπλέκει τα πράγματα στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συστήματος. Ναι, μπορεί, αλλά ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ας το προσπαθήσουμε. Υπάρχει τώρα ένα σημείο, το 16 αν δεν κάνω λάθος ή κάποιο άλλο, όπου εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τις ε, διασκέψεις εκείνες τις οποίες καλούνται μόνο κάποια εθνικά κοινοβούλια και όχι όλα. Η ενισχυμένη αυτή συνεργασία την οποία προωθώ με την έκθεσή μου θα πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για τις μελλοντικές διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτές οι διασκέψεις να έχουν περιορισμένη σύνθεση. Ακόμα και στις συνεδριάσεις αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας θα πρέπει η συμμετοχή των υπολείπων εθνικών κοινοβουλίων να προβλέπεται. Αν τώρα υπάρχουν κάποια εθνικά κοινοβούλια τα οποία θέλουν να βρεθούν μεταξύ τους με μικρή ας πούμε περιορισμένη σύνθεση δεν θα πρέπει να αποκλείουν στις συνεδριάσεις αυτές τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Μπορούν να συγκαλούν αν θέλουν τις διασκέψεις αυτές, αλλά να τις καθιστούν ανοιχτέ προς τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή τη διευκρίνηση ήθελα να δώσω. Λοιπόν, όσον αφορά τις τροπολογίες τώρα, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ξέρετε, επομένω θα πρέπει να προβλεφθεί αρκετά σύντομα, γιατί τελειώνει και αυτή η κοινοβουλευτική θητεία 17 Φεβρουαρίου 17 Φεβρουαρίου θα είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση το Μάρτιο. Κύριε Ντάφη, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω απολύτως ότι θέλετε να προχωρήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά η 17η του μήνα είναι η Δευτέρα της μεθεπόμενης εβδομάδας. Της επόμενης εβδομάδας. Και αν ως ομάδα θέλουμε να ανταποκριθούμε στην πολυπλοκότητα της έκθεσης αυτής, την οποία θα ήθελα να ξανατονίσω, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Φοβάμαι ότι εάν πιεστούμε να υποβάλουμε τροπολογίες μέσα σε μία εβδομάδα, δεν ε, θα ανταποκρίνονται στην ποιότητα που χρειαζόμαστε για την έκθεση αυτή. Κύριε Ντάφα, κοιτάξτε, πρέπει η έκθεση αυτή να πάει στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Άρα το Μάρτιο, το αργότερο, πρέπει να καταφέρουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και θα πρέπει προφανώς να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες. Τότε συμφωνείτε με την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε προθεσμία δύο εβδομάδων για να καταθέσουμε τροπολογίες. Io, però eh, Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινή, η γραμματεία μου λέει 20 Φεβρουαρίου ω μέση λύση. Συμφωνώ πάντως με την παρατήρησή σας κύριε Ντάφα. Είναι πολύ σημαντικό οι τροπολογίες αυτές να είναι καλής ποιότητος, να τις έχετε μελετήσει και να λύσει καλά, να είναι καλά διατυπωμένες και αυτό θα διευκολύνει το έργο μας. Ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σας κύριε Ντάφ, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Εγώ θα δεχόμουν τις 24 Φεβρουαρίου, η γραμματεία μου λέει 20 Φεβρουαρίου καλύτερα. Κερδίζουμε πάλι κάποιες μέρες και με αυτό. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά α κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να αποκριθούμε σε αυτή την προθεσμία. Κύριε Ντάφε, μένετε εσεί στην δική σα την πρόταση 24 Φεβρουαρίου. Ο κύριο Μορέιρα τι έχει να πει. Θα συμφωνούσα ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Είναι σημαντικό το θέμα, χρειαζόμαστε μια καλή έκθεση. Πολύ ωραία. 24 Φεβρουαρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 24 Φεβρουαρίου μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Και κάνω μια έκκληση να μην υποβάλλετε 300 ταυτόσιμες τροπολογίες, λίγες ευσύνοπτες ξεκάθαρες τροπολογίες. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε πλήρως και να τις εντάξουμε έπειτα στο κείμενο. Ε, με ενημέρωσαν για το υπόλοιπο της συνεδρίασης ότι ο κύριος Ράγγελ, ο οποίος θα παρουσίαζε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται ακόμα στη Λισαβόν εξαιτία κακοκαιρία. Θα αποχωρήσει, θα αναχωρήσει μάλλον του με δύο ώρες καθυστέρηση. Επομένως, ε, δεν θα φτάσει τουλάχιστον στην ώρα του, κάποια στιγμή αργότερα φανταζόμαστε. Όσον αφορά τώρα την έκθεση Σόλτς. Δεν έχουμε τους κοιόδης συγητές ακόμα. Φτάνουνε οι σκιώδεις ηγητές. Λοιπόν, να ζητήσω από τον κύριο Ντάφ τότε, αν είναι δυνατόν να... Λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Ραντζέλα θα καθυστερήσει και οι σκιώδεις ηγητές για την έκθεση Σόλτς δεν έχουν φτάσει ακόμα. Επομένως, Μπορούμε να συζητήσουμε πρώτα το σημείο 8 του κύριου Ντάφα. Συμφωνείτε κύριε Ντάφα. Κατά αυτόν τον τρόπο διευθετούμε και το πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα. Σας ζητώ, αντί να συζητήσουμε το σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, για την εργασία της Τρόικας και να συζητήσουμε το σημείο 6 ή και το 7, να περάσουμε μέσα στο σημείο 8 διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, διδάγματα που πρέπει να αντιληφθούν και μελλοντικές προοπτικές. Εσείς κύριε Ντάφη είστε συντάκτης γνωμοδότησης. Σας διορίσαμε στις 17 Δεκεμβρίου συντάκτη γνωμοδότησης και υποβάλλουμε στα πλαίσια του άρθρου 50 ως συνδεδεμένη επιτροπή τη γνωμοδότησή μας αυτή στην Επιτροπή Προπολογισμών. Αν συμφωνείτε λοιπόν και εσείς κύριε Ντάφα, κάντε τώρα την παρουσίασή σας. Ε, ε, um, Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, η σε γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιομικό πλαίσιο και τις αντίστοιχε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις ε, αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής ε, Προπολογισμών. Μίλησα ε, στους συνεισηγητές, τον κύριο Ντέν και τον κύριο Κάλφιν και σε γενικές γραμμές ε, στηρίζω την προσέγγιση τους. Η ευθύνη της ε, δικής μας επιτροπή είναι να εξετάσει την χρήση της ε, συνθήκης κατά τη διάρκεια των, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και των ίδιων πόρων. Έτσι ώστε να διαπιστώσουμε το πώς εφαρμόστηκαν οι διαδικαστικοί μας κανόνες. Με αυτόν τον ε, τρόπο έχουμε το βλέμμα στραμμένο τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα ξεκινήσει, βασικά έχει ήδη ξεκινήσει ε, δεδομένου ότι δημιουργήθηκε μια ομάδα μελέτης μόλις πριν από λίγο, ομάδα εργασίας, αλλά θα ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει το 2016. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο και στην ενδιάμεση έκθεση, αλλά και σε περαιτέρω τροποποίηση της ε, συνθήκης που είναι ενδεχομένως απαραίτητες ή επιθυμητές ή και τα δύο. προκειμένου να συμπληρωθεί η έκθεση Dean Calvin. Οι προτάσεις που σας υποβάλλω ως τροπολογίες ε, μπορώ να σας ε, πω ότι ήδη βρίσκουν σε γενικές γραμμές σύμφωνο τόσο των κύριο Ντεάν όσο και τον κύριο Κάλφιν. Ε, παρακολούθησα μια συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και το συζητήσαμε ήδη. Η επόμενη συνάντησή τους θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και θα παραστώ και πάλι. Αυτά ε, καταρχήν. Τώρα, ε, συνοπτικά για το τι προτείνω. Ε, θεωρώ ότι η Επιτροπή Σούρε, η οποία συστάθηκε ακριβώς ε, για να καθοριστεί και να προωθηθεί η άποψη του Κοινοβουλίου, ήταν ε, πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή. Η ιδέα της σύστασης ήταν πολύ καλή. τα συμπεράσματά της ήταν πολύ θετικά. Το θέμα είναι το κατά πόσον μπορέσαμε τα συμπεράσματα αυτά να τα προωθήσουμε στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά βάση κατέβασε τα ρολά μπροστά σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση των πολιτικών προτεραιοτήτων στη διάρκεια της οποίας θα μπορούσαμε να είχαμε επιμείνει και να είχαμε προβάλλει τα συμπεράσματα αυτά, για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά το ε, ύψος του προϋπολογισμού. Το περιθώριο ελιγμών μας ήταν ε, πολύ περιορισμένο σε ό,τι αφορά την διεύρυνση της διαπραγμάτευσης σε άλλα θέματα ε, κάτι που θα μας έδινε μια ευελιξία σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα. Στην τροπολογία μου μόνο 4 για την παράφορα 14 υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει δεν ασκεί νομοθετική εξουσία σύμφωνα με τη συνθήκη. και κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης κατά κάποιο τρόπο καταχράστηκε αρμοδιότητες. Στην τροπολογία μου μόνο έξι από την άλλη μεριά. Λέω ότι οι ε, ενδιάμεσες ε, διατάξεις που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο του Συμβουλίου και να επιταχύνουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Πέραν αυτού δε, καμία από τις προεδρίες αλλά ούτε και η Κομισιόν καν πρότειναν τη χρήση τους. Είτε της ε, γενικής ε, ενδιάμεσης διάταξης ούτε τις ειδικές ε, διατάξεις του άρθρου 212. που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να διευκολυνθεί η ε, λήξη των διαπραγματεύσεων και η ανέβρεση λύσης. Η έλλειψη ευελιξίας από πλευράς του, του Συμβουλίου Ε, ενίσχυσε τις ε, απόψεις περί ε, δίκαιης ανταμοιβής ή δίκαιου, δίκαιου ανταλλάγματος. Θυμάστε πόσο η κυρία Θάτσερ είχε υποστηρίξει αυτή την αρχή. Νομίζω ότι επισκίασε κατά κάποιο τρόπο τις διαπραγματεύσεις. Αναμένοντας λοιπόν την ενδιάμεση αξιολόγηση, Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες, τις ενδεχόμενες αδυναμίες της ε, ισχύουσας συμφωνίας. Μεταξύ αυτών που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει διάρκεια μικρότερη των 7 ετών. Το αναφέρω στην πρόταση τροπολογίας μου υπαριθμών 7. Το προσχέδιο της Επιτροπή, έκθεσης της Επιτροπής Προπολογισμών ε, ε, δεν ήταν πολύ σαφές για αυτό το θέμα. Εγώ επιμένω λοιπόν και Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις επόμενες διαπραγματεύσεις, όχι μόνο επειδή το επιτάσσει η δημοκρατία, αλλά και επειδή οι αποφάσεις για τις δαπάνες στο μέλλον θα απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Μετά στον εσωτερικό μας κανονισμό αναφέρουμε σε μια μάλλον σε μια συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρουμε στον εσωτερικό μας κανονισμό και συγκεκριμένα σε πέντε άρθρα του. δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη λογική συνέπεια, διότι έχουμε τροποποιήσει ε, το άρθρο 17α του εσωτερικού μας κανονισμού, το 17 και το 17α συγκεκριμένα, ε, που είναι τα άρθρα τα οποία πραγματικά θα ε, χρησιμοποιηθούν και θα αποτελέσουν το γνώμονα για τις επόμενες διαπραγματεύσεις για το λέτε νομικό πλαίσιο. Πάντως ε, αυτά τα άρθρα είναι σημαντικά για όλους τους εμπλεκόμενους στις διαπραγματεύσεις. Ε, δεύτερον, αναφέρομαι στον ρόλο του Προέδρου του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να τη σεβασμού αλλά και να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και τρίτον, ε, ε, αναφέρομαι στις σε ορισμένες ομάδες μειονότητες οι οποίες αποκλείστηκαν από την συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, αναφέρομαι στο κείμενό μου στις ε, απαραίτητες τροποποίησεις της συνθήκης. Λέω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αυθεντική ε, συναπόφαση εμείς με το, με το Συμβούλιο. Δεν αναφέρω λεπτομέρειε για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι ο γενικότερος χαρακτήρας της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι πιο δημοκρατικός, ε, θα πρέπει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να βρίσκονται στο, στο ίδιο επίπεδο ε, και ε, να μην υπερέχει το ένα το άλλο. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο. Κανείς λοιπόν δεν θέλει να πάρει το λόγο. Άρα ας καθαρίσουμε την... Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Προπολογισμών μέχρι τις 18 Μαρτίου πρέπει να υιοθετήσει την έκθεσή της. Άρα, εμείς πρέπει να καθορίσουμε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, τι να πούμε, 20 Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου συμφωνείτε, ή 24 Φεβρουαρίου, 20 Μπορείτε να δεχτείτε αυτή τη φορά την 20 Φεβρουαρίου ως ημερομηνία Κατάθεση τροπολογιών, πολύ ωραία. 12 το μεσημέρι. Θα προχωρήσουμε έτσι λοιπόν. 5. Allora, in attesa che arrivi il collega Rangel, il quale... Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα τον κύριο Ραντζέλ, ο οποίος έχει φτάσει στις Βρυξέλλες, δεν έχει φτάσει ακόμα στο Κοινοβούλιο. Περιμένοντάς το λοιπόν, σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, διερευνητική έκθεση για το ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην τελευταία μας συνεδρίαση, 21 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, συζητήσαμε το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσίασε ο κύριος Σόλτς. Έλαβε χώρα μια συζήτηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Κατατέθηκαν 37 τροπολογίε από τους Ραντζέλ, Σέπφλιν, Δρούτσα, Ντάφα, και από τον κύριο Σόλτ τον εισηγητή μας. Κύριε Σόλτ, πείτε μα ποια είναι η υποψή σα τώρα για τι τροπολογίε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέρφους που επεξεργάστηκαν τόσο βραχυπρόθεσμα το θέμα αυτό και έχουν υποβάλει τροπολογίες. Η καταπολέμηση της ε, κρίσης ε, και η εξελίξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κεντρικό θέμα για, την για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό δεν θα εκπλήξει και κανέναν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος της θητείας εξετάζει πώς έχουν διεξαθεί οι σχετικές εργασίες, ε, τι έχουν αποφέρει και όπως λέει και ο συνάδελφος Ράγγελ σε μία ε, τροπολογία του να εξάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ως Επιτροπή γνωμοδοτούμε για την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και ο συνάδελφο Κάραξ και ο Χουαν Κόκ, που είναι οι συγκητέ εκθέσεις, έχουν λάβει πάρα πολλέ τροπολογίε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και στην Επιτροπή ε, επί της ουσίας θεωρείται πολύ σημαντικό το θέμα. 37 ε, τροπολογίες έχουν υποβληθεί, τις έχω εξετάσει προσεκτικά και θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μένα. Και τα έχω συζητήσει ήδη με τους κοιόδης εισηγητές. Καταρχάς, Πιστεύω ότι με βάση τις τροπολογίες αυτές θα μπορέσουμε να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση την οποία ελπίζω θα μπορέσουν να στηρίξουν πολλοί συνάδελφοι και επίσης ε, κάτι που συνδέεται με το πρώτο θέμα. Ε, κανένας συνάδελφος δεν αμφισβητεί την ε, δομή και την προσέγγιση στο θέμα. Προσπάθησα να δείξω ότι... Ε, Προσπάθησα να δείξω πώς έχουν αντιδράσει τα θεσμικά όργανα ε, στην κρίση και με ποιες ε, νομικές βάσεις. Έχω εκπονήσει κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις, τις οποίες θα ήθελα σύντομα να παρουσιάσω. Καταρχάς έχουμε την λύση ad hoc, η οποία πριν κάποια χρόνια ε, αντικαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Σταθερότητας. Ε, τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ε, απειλεί να αυτονομηθεί. Θα θέλαμε λοιπόν εδώ μια τροποποίηση γιατί, διότι με βάση των οικονομικών αναγκών και με βάση την συνθήκη της Λισαβόνας είδαμε μια τρομερή κρίση στην ε, Ευρωζώνη και δημιουργήθηκε έτσι ένας ε, μηχανισμός ε, σταθεροποίησης από τον οποίο όμως απορρέουν φυγοκεντρικές δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση που ασχολείται αναλυτικά με τις ενέργειες της Τρόικας και που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Κοινοβούλιο. Στην γνωμοδότησή μου κάνω έκκληση οι δύο παράλληλοι μηχανισμοί που υπάρχουν για την Ευρωζώνη και για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης ε, να επανεξεταστούν και Υποθέτω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε κι εσείς ε, αυτήν ε, την προσέγγιση. Στο άρθρο 143 της συνθήκης ε, υπάρχει μία δυνατότητα Ε, παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Δεύτερον, οι ενέργειες ε, των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ε, τη Τρόικα, ε, του μηχανισμού σταθεροποίησης δηλαδή, δεν υπόκεινται σε υποχρέωση λογοδοσίας και το θέμα αυτό δεν τίθεται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά Φαίνεται και στην έκθεση κάρα Κενγκόκ ότι ότι ε, ε, υπάρχει ε, διαδικασία συναπόφασης όσον αφορά τις προϋποθέσεις αλλά αυτό δεν αποτελεί το επίκεντρο της δικής μας γνωμοδότησης. Πολιτικά θα πρέπει στην Επιτροπή μας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο πλαίσιο των φόρουμ συνεργασίας που υπάρχουν. Και κύριε Πρόεδρε, και εσείς στην έκθεσή σας ασχοληθήκατε με τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Τρίτον, στις ε, τροπολογίες κατά τη γνώμη μου φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τα μνημόνια που ε, εκπώνησε η Τρόικα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές συνέπειες και τα μέτρα θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δηλαδή την οικονομική σταθερότητα, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, κοινωνική σταθερότητα στα κράτη-μέλη. Το τελευταίο αυτό συνδέεται και με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι πολύ σημαντικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα που ενεργούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Αυτό το θέμα όμως δεν αποτελεί επίκεντρο για τη δική μας Επιτροπή. Θεωρώ τέλος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στα θέματα αυτά να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό από τον οποίο να απορρέει ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τίθενται λοιπόν πολλά ερωτήματα σχετικά με την άσκηση των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει τα όρια της εκθέσης αυτής, θα πρέπει όμως να τονιστεί σε πολιτικό πλαίσιο. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις των σχεδόν εισαγητητών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σόλτ, Έχουμε ήδη ένα κατάλογο μιλητών. Ο κύριος Μπρόκ πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συμφωνήσω όσον αφορά τα θεσμικά θέματα. Αυτά έχουν συζητηθεί και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Το Συμβούλιο, η Προεδρία της Ευρωζώνης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και η Κομισιόν έχουν εξηγήσει ότι θα πρέπει ο μηχανισμός σταθερότητας ε, να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο όσο γίνεται πιο σύντομα. υπάρχει αυτή η υποχρέωση των θεσμικών οργάνων απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Εμένα όμως ε, μου λείπουν δύο πράγματα ως προς το περιεχόμενο καταρχάς. Ε, όλο το φταίξιμο εδώ πέρα ρίχνεται στην Τρόικα και στη διαδικασία. Αλλά η κατάσταση κάποιων κρατών μελών οφείλεται και σε λάθη που έγιναν εντός των κρατών μελών. Αλλιώς δεν θα είχαν φτάσει ποτέ στην κρίση να θεωρούμε την Τρόικα υπεύθυνη για την, ε, για την κρίση μου φαίνεται υπερβολικό. Εάν τα κράτη-μέλη αυτά είχαν ρυθμίσει καλύτερα το τραπεζικό του σύστημα, εάν είχαν καλύτερη ανταγωνιστικότητα, δεν θα είχαν καταλήξει ε, ποτέ σε αυτήν την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή την ιδέα θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε. Το θέμα ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας οδηγεί σε προβλήματα στην αγορά εργασίας δεν ε, σχετίζεται με τα μέτρα που ε, αναγκάστηκε να λάβει η Τρόικα. Η Τρόικα εμπόδισε να ε, φτάσουν τα κράτη αυτά σε αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά την αποπληρωμή των χρεών. Επίσης, Ε, όσον αφορά ε, τη στρατηγική 2020. Οι στρατηγικές αυτές έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Επειδή δεν ήταν ανταγωνιστικά, βρέθηκαν στην κρίση. Δεν έχουν εφαρμόσει τη στρατηγική αυτή σωστή. Αυτό όμως δεν μπορούμε ε, να θεωρήσουμε ότι είναι φταίξιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέτρα που θα έπρεπε να έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ ε, πιστεύω ότι λείπουν κάποιες αποχρώσεις, για να το πω ευγενικά. Και επίσης οι συνέπειες μιας έλλειψης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σημαίνει ότι ε, θα μπορούσαν να συνεχίζουν να γίνονται πληρωμές ε, κοινωνικής ασφάλειας ε, στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι μάλλον θα μπορούσε να συνεχίσει να γίνεται αυτό εάν δεν δινόντουσαν ευρωπαϊκές πληρωμές στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να πληρωθεί κανένας μισθός, καμία σύνταξη. Διότι το ίδιο το κράτος δεν θα μπορούσε να πληρώσει τα χρήματα αυτά. και πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη εάν θέλουμε να φτάσουμε σε κάποια δίκαιη αξιολόγηση της κατάστασης. Πριν 1,5 χρόνο βρέθηκα στην Ελλάδα. Τότε που ανέλαβε την κυβέρνηση ο, ο Σαμαράς. Και μίλησα τότε με ε, την... Ε, με την ε, διοίκηση του, των κοινωνικών εταίρων. Αλλά δεν έγινε καμία συζήτηση ανάμεσα στην κυβέρνηση, ε, τους εργοδότες ε, και εργαζομένων. Αυτό όμως δεν είναι λάθος της Τρόικας, είναι λάθος της κρατικής πολιτικής. Και αυτό ισχύει και για άλλα κράτη-μέλη που έχουν την παράδοση των κοινωνικών εταίρων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό ή να αφαιρέσουμε τελείω ε, την ε, πολιτική αξιολόγηση. Η πολιτική αξιολόγηση που υπάρχει εδώ πέρα δεν είναι σωστή, δεν είναι δίκαιη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, και τα θέματα αυτά. Να αφαιρέσουμε δηλαδή την ιδεολογική αξιολόγηση και να επικεντρωθούμε στα θεσμικά θέματα, στα οποία σύντομα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση. Και αν αφαιρέσουμε τα άλλα αυτά σημεία, σύντομα θα συμφωνήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε στη γνωμοδότηση αυτή να κάνουμε οι οικονομικοπολιτικές επικρίσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τις εργασίες ε, της Επιτροπής μας. Συγγνώμη, πρέπει σε πέντε λεπτά να αποχωρήσω γιατί πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Ζητώ από την κυρία Λεγκρίπ αν μπορεί να αναλάβει λίγο την Προεδρία μέχρι να επιστρέψω. Ρέντνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής ε, των Σοσιαλδημοκρατών ε, λείπει λόγω ασθενείας. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σόλτς για τον τρόπο με τον οποίο έχει διατυπώσει τη γνωμοδότηση αυτή και με τον τρόπο που έχει, για τον τρόπο που έχει συνεργαστεί με τους σκιώδεις συζητητές... και όσον αφορά το περιεχόμενο. Πιο σημαντικό είναι το επίκεντρο στο, στην συμβολή που μπορεί να έχει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Πρέπει να έχουμε ευρία οπτική Ωστόσο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι αρμοδιότητες στο θέμα αυτό. Η τρόικα αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί από ε, μια νομικά αιτιολογημένη δομή, κάτι που να, είναι, που να έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση. Όλα τα προβλήματα επί του περιεχομένου που ανέφερε και ο συνάδελφος Μπροκ μπορούν ε, ε, να έχουν ε, οδηγήσει στα προβλήματα και ο κύριος Μπροκ λείπει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να αναφέρω το εξή που ανέφερε και εκείνο. Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση ε, και όσον αφορά τους στόχους 2020, το θέμα εδώ δεν είναι ε, η ανταγωνιστικότητα, ναι, αλλά το θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Και θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το συνολικό αυτό πακέτο και γι' αυτό οι συστάσεις αυτές ε, είναι απόλυτα αιτιολογημένε και πολύ καλά διατυπωμένε. Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση που ε, ανέφερε και ο συνάδελφο Σόλ είναι η αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είπε σήμερα ο Ότμαρ Καράς, ε, αλλά αναφέρθηκε στη, στο δημοψήφισμα στην Ελβετία, δεν είναι από το σούσι που διαλέγουμε από την κορδέλα που περνάει είναι θεμελιώδη δικαιώματα και ε, έχουμε την ε, νομική αξιολόγηση του ε, καθηγητή Φυσελεσκάνο, ένα μνημόνιο κατανόησης δεν επιτρέπεται να παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Θα πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον να μην ε, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτά λοιπόν είναι τα, συνα... τα μηνύματα του συναδέλφου Τούτσα. Ο λόγος του κύριου Νταφ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως υπάρχουν δύο πράγματα που δεν μπορώ να υποστηρίξω. Πρώτον, η πρώτη. Υπονοείται ότι η Τρόικα δεν έχει νομιμοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Υπό, δεν έχει νομιμοποίηση υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τουλάχιστον. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά ακόμα και αν ήταν σωστό, ακόμα και αν ήταν, μάλλον αν ήταν αληθές, θα βρισκόμασταν σε πάρα πολύ δυσχερή πολιτικά και νομικά θέση. Το καθήκον της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ε, Κομισιόν είναι να μεριμνούν έτσι ώστε το ευρώ να είναι ένα νόμισμα όσο πιο σταθερό γίνεται. Και επίσης να μεριμνούν έτσι ώστε να υφίστανται οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ε, ε οικονομική ε, ανόρθωση. Αυτό απαιτεί από ορισμένε τουλάχιστον χώρε σημαντικές διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανωμένες και τη αγορά εργασίας. Και μάλιστα επίσης απαιτεί να δοθεί ένα τέλος στις απάτες που στην Ιρλανδία και την Ελλάδα είχαν φτάσει σε ε, επικίνδυνα υψηλό ποσοστό. Και η Τρόικα πετυχαίνει ε, το στόχο της ε, εξασφάλισης πιο σωστών συνθήκων σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε, όπως είπε ο κύριος Μπροκ, το, το πρόγραμμα, τα προγράμματα της Τρόικας στο σύνολό τους, όχι μόνο να εντοπίζουμε κάποιες πτυχές τους τις οποίες δεν θεωρούμε επιθυμητές. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ότι ε, απέτυχε να διορθώσει τις ε, ε, τη νομική βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η δημιουργία της Τρόικα. Καλέσαμε το Συμβούλιο να δημιουργήσει μέσω της τροπής των συνθήκων ε, ένα διαφορετικό, ένα διαφορετικό σύνολο από κανόνες αλλά γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα της Τρόικα ε, είναι επίγουσας εφαρμογής, δηλαδή είναι προσωρινά προγράμματα εν ώψη μιας κρίσης. Δεν θα διαρκέσουν για πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι έχουν νομιμοποίηση και στόχο και λόγο ύπαρξης. δίνουν και αποτελέσματα. Βέβαια, υπάρχουν και συνέπειες και είναι σημαντικό να πούμε ως Κοινοβούλιο ότι έχουμε συνείδηση αυτών των συνεπειών, ότι ανησυχούμε για τις κοινωνικές ιδιαίτερους συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Όμως, επίσης πιστεύω ότι δεν θα πρέπει ε, να δημιουργούμε θεμελιώδη δικαιώματα εκ του μειόντος. Η χάρτα των θεμελιών δικαιωμάτων έχει δύο τύπους διατάξεων. Τα κλασικά θεμελιώδη δικαιώματα και τις κοινωνικές αρχές. Εδώ μιλούμε για κοινωνικές αρχές και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτών και των κλασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το να επικαλούμαστε τη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υποστηρίξουμε τις επικρίσεις μας προς το Συμβούλιο, όπως κάνει η έκθεση, νομίζω ότι μερικές φορές απαξιώνει τη χάρτα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβαστική πρόταση J που διακρίνει το ρόλο του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και δίνει ηγετικό ρόλο στην Κομισιόν τόσο στην Τρόικα όσο και στο όργανο που θα πρέπει να λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, η συμβαστική πρόταση D δεν νομίζω ότι είναι ορθή. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να λέμε ότι η διαδικασία ε, διακεί υπερβολικά. Ήταν εξ αρχής σαφές ότι οι διαστοτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες ζήτησε η Τρόικα δεν, μπορούν να, δεν μπορούσαν να δώσουν μια ε, άμεση απάντηση στην κρίση. Θα πάρει χρόνο, δεκαετίες ολόκληρες, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως και να δώσουν τα πλήρη αποτελέσματά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πάολο Ράγγελ. Πάολο Ράγγελ, μάλλον, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτς για την ε, συμβαστικές του προτάσεις. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο, μάλλον σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει, αλλά υπάρχουν, αν μη τι άλλο, δύο ή τρεις συμβαστικές προτάσεις οι οποίες ακόμα και αν προσπαθούν να συμπεριλάβουν κάπως την προτινόμενη από μένα διατύπωση και όντως το κάνουν αυτό, παρόλα αυτά δεν συνάδουν με το πνεύμα των προτάσεών μου. Ουσιαστικά, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Προέρχομαι από μια χώρα όπου είχαμε και έχουμε ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιβληθεί από την Τρόικα. Επομένως, έχουμε ήδη μια κάποια εμπειρία του τι σημαίνει να υπάγεται κανείς σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι έχουμε τώρα ενώπιόν μας όχι μόνο την γνωμοδότηση αυτή, αλλά και την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. η οποία και αυτή έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα σε ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο της μέρος. Ενώπιον μας λοιπόν έχουμε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση. Δεν λέω ότι είναι λάθος αυτό, απλώς θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Στην συμβαστική πρόταση C για παράδειγμα, έλεγα ότι δεν υφίσταται, δεν έλεγα ότι δεν υφίσταται ένας κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος. Λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρξει ένας δημοκρατικός έλεγχος, να προβλέπεται δημοκρατικός έλεγχος. Σε μια δική μου τροπολογία λέω κάτι τέτοιο. Ας μην ξεχνάμε ότι σε κάθε χώρα που είχαμε παρούσα την Τρόικα, έλαβαν χώρα και εθνικές εκλογές, όπου μια μεγάλη πλειοψηφία κατά κάποιο τρόπο επικύρωσε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι εγκρίθηκε ξεχωριστά κάθε διάταξη του μνημονίου αυτού αν θέλετε, εγκρίθηκαν οι γενικότερες κατευθύνες γραμμές που προέβλεπαν πολιτική λιτότητος, θυσίες και πολύ αυστηρά μέτρα. Όλα αυτά γίνουν αποδεκτά ως μία λύση για την κατεπίγουσα αυτή κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι χώρες αυτές. Θυμάμαι ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου με την Ιρλανδία γίνουν εθνικές εκλογές, μετά την υπογραφή του μνημονίου της Πορτογαλίας ακολούθησαν εθνικές εκλογές Κατά τη διάρκεια της υπογραφής του δεύτερου μνημονίου γίνανε δύο φορές εκλογές και δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι η αλλαγή του Προέδρου στην Κύπρο ουσιαστικά συνέπεσε πάνω κάτω με την υπογραφή του μνημονίου. Όταν μιλάμε λοιπόν για δημοκρατικό έλλειμμα, αναφερόμαθα όχι μόνο στις μη στις συζητήσεις που δεν γίνανε στα κοινοβούλια, αναφερόμαστε ολότελα σε εθνικές εκλογές οι οποίες έλαβαν χώρα λίγο πριν ή μετά την υπογραφή των μνημονίων αυτών. Εντάξει, δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι ήταν μη δημοκρατική η μετα την υπογραφη των μνημονιων αυτων δεν μπορουμε λοιπον να λεμε οτι ηταν μη δημοκρατικη η κατασταση τη στιγμή που γίνανε εθνικές εκλογές, σε ένα 80% των ψηφοφόρων στην Πορτογαλία τάχθηκαν υπέρ πολιτικών κομμάτων που επισήμως είχαν υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης και 90% των βουλευτών του Εθνικού μας Κοινοβουλίου ουσιαστικά ενέκριναν το μνημόνιο αυτό και είχαμε εκλογέ μετά από ένα μήνα στην Πορτογαλία και αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στην Ιρλανδία. Αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή είναι το να προωθούμε μια θεωρία όπου λέμε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά δημοκρατική βούληση στην όλη αυτή τη δικασία, προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό. Μπορούμε προφανώς να πούμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία υπερβαίνουν για παράδειγμα το μνημόνιο αυτό ή κάποια μέτρα τα οποία δεν θα δεχόταν εύκολα ο λαός. Οι γενικές πάντως κατευθύνες γραμμές εγκρίθηκαν όχι μόνο μέσω κοινοβουλίων, αλλά μέσω εθνικών εκλογών. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριο Μπρόκ, να καταφέρουμε να περιορίσουμε την γνωμοδότησή μα στα θεσμικά μόνο ζητήματα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό μηχανισμό που να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια τέτοια οικονομική κρίση ενδεχομένως θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια νέα θεσμική ερτεκτονική στο μέλλον προκειμένου να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει, για παράδειγμα, με την Τραπεζική Ένωση, όχι όπως προτείνεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο, αλλά όπως ουσιαστικά θέλει να τη δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή λύση για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιες κρίσεις όπως είδαμε στην Κύπρο, στην Ιρλανδία ή την Ισπανία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο για μένα. Πάντως, στη συμβαστική πρόταση Γ θεωρώ ότι είναι κάπως υπερβολικό να λέμε τα όσα λέμε. Το ίδιο ισχύει και για τη συμβαστική πρόταση G, η οποία πραγματικά δεν αποτελεί συμβιβασμό και νομίζω ότι αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και συμβαστική πρόταση I. Πρέπει βέβαια να πω ότι έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες από το συντάκτη γνωμοδότησης, όπου την αρχική του πρόταση έχουμε φτάσει σε αυτούς τους σημαντικούς συμβιβασμούς. Καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι έχετε καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες για να συγκεράσετε τις διάφορες απόψεις. Ωστόσο πρέπει να πω ότι κατά τη δική μου την άποψη δεν αρκεί να χρησιμοποιούμε απλώς ή να χρησιμοποιείτε εσείς κάποιες δικές μας διατυπώσεις και εκφράσεις και να θεωρείτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε σε συμβασμό. Το θέμα δεν είναι η διατύπωση, το θέμα είναι η πρόθεση που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Για παράδειγμα, συμβαστική πρόταση Γ δεν νομίζω ότι εκτοπτρίζεται η αρχική μου πρόθεση και το ίδιο συμβαίνει και η συμβαστική πρόταση G. Έχετε απλώς χρησιμοποιήσει κάποιες δικές μου εκφράσεις. Το γενικότερο όμως πνεύμα, η γενικότερη πρόθεση των προτάσεών μου δεν αντικατοπτρίζεται στην συμβαστική πρόταση. Πολλές φορές λέει ακριβώς το αντίθετο. Θα ήταν πιο σκόπιμο λοιπόν να περιοριστούμε περισσότερο στα θεσμικά ζητήματα, στη θεσμική πτυχή της γνωμοδότησης, επί της οποίας άλλωστε συμφωνούμε ως επιτοπλίστων, και στη τελευταία ανάρτηση, εμεί δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδια επιτροπή αυτή τη στιγμή. Είμαστε επιτροπή σταγματικών υποθέσεων που γνωμοδοτεί, άρα επί των ε, θεσμικών ζητημάτων πρέπει να τοποθετηθούμε και όχι επί των ιδεολογικών θεμάτων. Είχα υποβάλει επίση και κάποιε τροπολογίε, γιατί θεωρώ ότι ακόμα και η έκθεση τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων απομακρύνεται κάπω από του βασικού αυτού κύριου στόχου. Ιδίω όταν ουσιαστικά ξεχνάει ότι έλαβαν χώρα, το παραλαμβάνω, εθνικές εκλογές σε κάθε χώρα που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Τρόικας. Έγιναν εθνικές εκλογές, ενώ υπήρχε πλήρης γνώση στη χώρα, στις χώρες εκείνες, του προγράμματος που πρότεινε η Τρόικα. Έγιναν εθνικές εκλογές αφού είχαν προηγηθεί πολύ έντονες βίες θαλασσιζητήσεις και ακόμα και στην Πορτογαλία, ακόμα και στην Κύπρο εγκρίθηκαν τα μνημόνια αυτά. Ξέρουμε ότι η κατάσταση δεν ήταν απόλυτα σαφή στην αρχή στην Ελλάδα με τις πρώτες εκλογές, ακολούθησαν και δεύτερες εκλογές, υπήρχε ένας κάποιο διχασμός, αλλά στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών ήταν σαφές. Θα μου πείτε βέβαια ότι πολλά άτομα, πολλοί άνθρωποι είναι κατά των μνημονίων αυτών. Είναι κατά όμως των μέτρων περισσότερο που βάλουν κυρίως κατά αυτών, κατά της δικής τους ομάδας. Όταν ρωτήσετε τους ανθρώπους αυτούς θέλετε να σώσετε τη χώρα από τη χροκοπία, λένε ναι και γνωρίζουμε ότι αυτό προποθέτει θυσίες. Όριμη λοιπόν η στάση των ανθρώπων απέναντι στα μνημόνια. Ας μην ξεχνάμε όμως και το νοσιακό επίπεδο, αλλά ας μην ξεχνάμε και το εθνικό είχαμε εθνικές εκλογές σε αυτές τις χώρες τι πιο δημοκρατικό από το να διοργανωθούν εθνικές εκλογές μετά την υπογραφή των μνημονίων. Και στη συνέχεια το αποτέλεσμα ήταν 80% των ψηφοφόρων ή των πολιτικών κομμάτων υπέρ των μνημονίων αυτών. Πώς μπορείτε να μιλάτε για δημοκρατικό έλλειμμα στη συνέχεια. Πώς μπορείτε να μιλάτε για απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης. Τι παραπάνω θέλετε, υπάρχει καλύτερη απόδειξη δημοκρατικής νομιμοποίησης από τις εκλογές. Μπορεί να μην σας αρέσουν τα μνημόνια αυτά. Ξέρετε, πολλές φορές ο άρρωστος θα πρέπει να αποδεχθεί και μια θεραπεία, ακόμα και πόδινη, προκειμένου να γίνει καλά. Μπορεί να μην σας αρέσει η θεραπεία, αλλά εν τέλει ξέρετε ότι πρέπει να υποστείτε αυτή τη θεραπεία. Λοιπόν, Να κάνω κι εγώ μια σύσταση λοιπόν με την άδειά σα. Α περιορίσουμε τι παρατηρήσει μα, τουλάχιστον εδώ στην Επιτροπή μα, στα θεσμικά μόνο ζητήματα, επί των οποίων εγώ συμφωνώ πλήρω με τη δική σα την προσέγγιση ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα θεσμικό μηχανισμό ανταπόκριση σε αυτέ τι κρίσει και ενδεχομένω να πρέπει να έχουμε και ένα θεσμικό μηχανισμό προληπτικό για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιε κρίσει, όχι μόνο για να τι επιλύουμε. Επ' αυτό νομίζω ότι έχουμε βρει ασυνένεση. Ωστόσο, θεωρούσα σημαντικό να πω ότι μολονότι έχουν υποβληθεί σημαντικότατες προσπάθειες για να καταλήξουμε στι συμβαστικές προτάσεις, έχω ουσιαστικέ αντιρρήσεις με πολλές από αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόλτ έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ θερμά για τις θέσεις των σκιωδών ε, εισηγητών αλλά και των συναδέφων από την Επιτροπή. Τρεις παρατηρήσεις είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικές στη συζήτηση αυτή. Αιτίες και αποτελέσματα. Μπορούμε να συζητούμε πολλή ώρα. Τι έφερε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέση αυτή αλλά μας ενδιαφέρει η νομική βάση, η δομή και η εντολή της Τρόικα, η δημοκρατική της νομιμοποίηση, η θεωρητική βάση για τις αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη στατιστικές, ε, οικονομικές προβλέψεις κλπ και στο πλαίσιο της έκθεσης ε, αλλά και των γνωμοδοτήσεων που πρόκειται να υποβάλουν και οι άλλες επιτροπές ε, πέρα από την ΑΦΚΟ, δηλαδή έχουμε την Επιτροπή Επασχόλησης, την Επιτροπή Χρηματο... Ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Νομικών Υποθέσεων και να εξετάσουμε τις συνέπειες. Εάν λοιπόν αυτό είναι το καθήκον μας, θα πρέπει εμείς ως Επιτροπή ΑΦΚΟ να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτά και να διαπιστώσουμε ότι με την Τρόικα εφαρμόστηκε μία πολιτική η οποία στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο δεν οδήγησε σε βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει λοιπόν να το κρίνουμε αυτό. Και Φυσικά είναι θέμα, της, είναι θέμα ιδεολογίας, αλλά είναι και θέμα αντίληψης ε, της πραγματικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τις κυβερνητικές δομές, τις ενέργειες ε, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να το αξιολογήσουμε αυτό και με τα μάτια της Επιτροπής μας. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνει κανείς ε, τις αιτίες και τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεύτερον, έχουμε το θέμα της νομιμοποίησης. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να τηρείται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως ε, να μιλάμε και για αποκατάσταση. Η απάντηση στα θέματα αυτά είναι πάντα πολύπλοκη και έχει να κάνει με την πραγματικότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε. Οι δυνάμεις μόχλευσης και μάλιστα όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα αλλά και από την Τρόικα. Όλες αυτές συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι την τελευταία προσφυγή στο συνταγματικό δίκαιο της Γερμανίας σχετικά με τα κρατικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι θέλουν να αποδείξουν με αυτήν την προσφυγή και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση σε δύσκολη οικονομική κατάσταση να αναπτύξει ένα μηχανισμό που να μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ξεπερνάσουν ε, την κρίση. Και μπορεί έτσι να διατηρηθεί και η υποστήριξη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως να μην διάβασα καλά το κείμενο, αλλά έχω την εντύπωση ότι στην ε, τροπολογία 8 Λέτε ότι απειλούνται τα κοινωνικά δικαιώματα των ε, πολιτών ε, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη δημοκρατική λογοθεσία. Την κατάλληλη την έχω υιοθετήσει κι εγώ. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε εμείς ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι δεν κατάλαβα το στόχο της τροπολογίας σας. Ε, προσπάθησα όμως ε, να την συμπεριλάβω σε μια συμβιβαστική τροπολογία. Κύριε Ράνιελ, και επίσης ε, στην τροπολογία 12 λέτε ότι στο εξή θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη προσέγγιση και ένα μηχανισμό που θα επικεντρώνονται στου στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προκειμένου να αποτρέπονται και να αντιμετωπίζονται παρόμοιε καταστάσει. Νομίζω ότι και εδώ τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω αυτό, νομίζω ότι και αυτή η τροπολογία σας έχει καλυφθεί από τη συμβαστική μου τροπολογία. Προσπαθώ ακριβώς αυτό το νόημα να συμπεριλάβω στο γενικό πλαίσιο. Γενικά λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό καθήκον της Επιτροπής μας να γνωμοδοτήσει. Ε, ήδη αναφέρθηκα στο πόσες τροπολογίες έχουν υποβληθεί στην ΕΚΟΝ Σημαντικό είναι λοιπόν με μια τέτοια γνωμοδότηση να υποδείξουμε έναν δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται καλύτερα σε καταστάσεις κρίσης και που να μπορεί να αποτελεί βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σόλτς. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε την εκθεσή σας από τις 10.30 και μετά. Έχουμε μία ώρα μόνο μπροστά μας ακόμα και πρέπει να καλύψουμε δύο σημαντικές εκθέσεις. Η πρώτη είναι η έκθεση του κύριου Ρανζέλ, σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνα ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα όμως τώρα. Μέχρι τις 6, 6 και 10 πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό για να αφιερώσουμε τα εναπομείναντα 20 λεπτά στην έκθεση της κυρίας Γκουρμάη. Το λόγο έχει ο κύριος Ρανζέλ. So, uh, Ευχαριστώ. Μια και ο χρόνος πιέζει, θα είμαι πολύ σύντομος. Δώσαμε το κείμενο ε, των ε, συμβαστικών προτάσεων, αλλά δεν ξέρω αν έχουν ήδη διανεμηθεί. Είναι το σχεδόν τελικό κείμενο, ναι μου λένε, ωραία. Έχω και εδώ μερικά αντίγραφα αν χρειάζεστε. Να πω το εξής. Λάβαμε πολλές ε, προτάσεις τροπολογίας. Οι πιο βασικές ιδέες ε, νομίζω μας βρίσκουν σύμφωνους όλους. Υπάρχουν όμως δύο-τρία επίμαχα θέματα για τα οποία εκφράστηκαν κάποιες διαφωνίες. έκανα προσπάθεια πραγματικά να συμπεριλάβω όλες τις οπτικές ε, του στις συμβαστικές μου προτάσεις. Πιστεύω ότι ακόμα και έτσι όμως ε, μπορούν να παραμείνουν κάποιες διαφωνίες. Σε αυτές θα εστιαστώ και όταν οι συνάδελφοι πάρουν το λόγο μπορούν επίσης να σχολιάσουν και να σχολιάσουν και άλλα ζητήματα ενδεχομένως. Ίσως υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη συμβαστική πρόταση F. Τι προσπάθησαμε να κάνουμε. Ε, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα της Κομισιόν και τις διάφορες δυνατότητες, διάφορες λύσεις. Προσπαθήσαμε να αφήσουμε ε, ανοιχτή μια λύση, έτσι ώστε να δώσουμε την ιδέα των clusters θεωρώντας ότι κάθε κλάση, σε κάθε κλάση θα προεδρεύει ένας αντιπρόεδρος, η σοσιαλιστική ομάδα το ζήτησε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε τέσσερις τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά κάνει ένα πρόβλημα. Και να αναφέρουμε επίσης και την ιδέα ότι στο μέλλον μπορούμε να έχουμε και επιτρόπους χωρίς χαρτοφυλάκιο. Αυτό δεν θα σημαίνει πως θα παραβούμε την, τον κανόνα του κάθε κράτος ε, ένας επίτροπος, ούτε την αρχή του κάθε επίτροπος μία ψήφος. Όχι. Θέλουμε να αφήσουμε τα διάφορα θερμικά όργανα να μπορούν να αυτοοργανωθούν. Και ο στόχος μας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου της Κομισιόν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κάποιον από αυτούς τους τρόπους. Κάποιο τύπο που είναι πολύ σημαντικό και επίμαχο ταυτόχρονα είναι επίσης το εξής. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την πλειοψηφία που χρειάζεται για μια πρόταση μομφής. Όμως, έχουν εκφραστεί δισταγμοί σε ό,τι αφορά την πρόταση, η πρόταση μορφής να απαιτεί απλή πλειοψηφία. Δηλαδή 376 ψήφους. Αυτή είναι η απλή πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου. Θα είναι η απλή πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ο συνάδελφος Ντάφ νομίζω πρότεινε να συμπεριλάβουμε και τη φράση χωρίς να διακινδυνεύσουμε, να θέσουμε σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις μορφής θα είναι επικοδομητικές. Όμως, δεν θα ήθελα ε, να ε, να υιοθετήσουμε ένα σύστημα που να μοιάζει τόσο πολύ με το γερμανικό και το ισπανικό. Θέλουμε το κοινοβούλιο να παίζει ένα ρόλο, αλλά όχι αυτός ο ρόλος της της, ε, όχι αυτή, ε, αυτός ρόλος να μην είναι η έννοια της επικοδομητικής πρότασης μορφής ακριβώς όπως την αναφέρει το γερμανικό ή το ισπανικό σύνταγμα. Επίσης, ένα άλλο θέμα, στο οποίο υπάρχουν κάποιες τριβές, προτάσεις Γκερέρο, ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα στην Κομισιόν, ότι θα προτείνουμε, θα υποβάλουμε ένα πρόγραμμα στην αρχή της θητείας της Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Όλα όσα προτείνω αποβλέπουν στην, στο διαχωρισμό των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι δικαιοδοσία της Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ασκεί εκτελεστική αρμοδιότητα. Θέλω η Κομισιόν να έχει τη δικαιοδοσία να ε, εγκρίνει το δικό της πρόγραμμα. Εμείς θα το επηρεάσουμε βέβαια και ήδη το κάνουμε. Το κάναμε. Το 2009 για παράδειγμα. Όταν αναβάλαμε την ψηφοφορία για τον πρόεδρο Μπαρόσο προκειμένου να τον υποχρεώσουμε να υποβάλει στο κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα και όπως γνωρίζουν ορισμένοι συνάδελφοι ο κύριος Μπαρόσο έκανε ένα πολύ δυναμικό θα έλεγα διάλογο τόσο με μέλη του Κοινοβουλίου όσο και με ολόκληρες επιτροπές πριν υποβάλει αυτό το πρόγραμμα. Συνεπώς ας αφήσουμε αυτό το θέμα στη δικαιοσία της Κομισιόν. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα αυτό της αυτονομίας της Κομισιόν και του Προέδρου της. Νομίζω ότι η πρόταση, τελευταία μας πρόταση ε, ευθυγραμμίζεται πιο πολύ και συμβαίνει πιο πολύ με αυτό πρότειναν νομίζω ορισμένοι βουλευτές του ΕΛΚ. Λέμε κατά βάση ότι για να είναι αποτελεσματική κομισιόν θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο όργανο. Όπερ σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν θα πρέπει να έχει στα χέρια του ε, εργαλεία οργάνωσης και πειθαρχία στην Κομισιόν. Αναγνωρίζουμε λοιπόν την αυτονομία του, συστήνουμε την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στα δύο φύλλα, και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Πρόεδρου της Κομισιόν να απορρίψει μια πρόταση κράτους μέλους για διορισμό επιτρόπου. Υπάρχει ήδη αυτό, αυτή η δυνατότητα, αλλά πρότεινα να διαγράψουμε, να μην δεχτούμε την πρόταση για τρεις ε, προϋποψηφίους. Το έχω διαγράψει αυτό το συμβασμό πια. Οπότε ανάμεσα στη συμβαστική πρόταση E, F, I και ίσως την όμικρον μάλλον με αυτές τις τροπολογίες ιδιαίτερως, ρυθμίζονται τα περισσότερα θέματα. Ελπίζω ότι οι επόμενες 18 ώρες θα είναι αρκετές για να επιλύσουμε και τα υπόλοιπα θεματάκια τα οποία μπορεί να παραμένουν. Είναι πραγματικά μικρές διαφορές οι οποίες παραμένουν αυτή τη στιγμή. Περιμένω τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας προκειμένου να βρούμε μια τελική συνένεση. Ευχαριστούμε κύριε Ραντζέλ. Ο κύριος Σέπλιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Πάολο Ραντζέλ. Θα είμαι πολύ σύντομος, ιδιαίτερα λακωνικός. Δεν είμαι ακόμα σαφώς υπέρ αυτής της ιδέας των επιτρόπων χωρίς χαρτοφυλάκιο. Ας το εξετάσουμε εκ νέου αυτό. Ουσιαστικά θα καταλήξει σε μία ανισότητα όσον αφορά το καθεστώς των επιτρόπων και ακριβώς αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Χρειαζόμαστε ισότητα των επιτρόπων για το σημείο ε, ισότητα των δύο Συμφωνούμε, clusters, αυτές οι ομάδες που βλέπουμε στην παράγραφο F, επί της αρχής μπορώ να συμφωνήσω. Θα θέλω όμως να γνωρίζω πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Δηλαδή, μπορεί στις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων να ταχθεί κανείς κατά των κλάστρες αυτών, σε ποιο σημείο της διαδικασία προβλέπονται, πότε μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει ότι θεωρούμε ότι δεν θα λειτουργήσει σωστά, πώς θα διοργανωθεί στην πράξη αυτή η διαδικασία. Αργότερα, στο σημείο H, αναφέρεστε στα αγγλικά στον όρο specificity, ιδιαιτερότητα. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό. Τουλάχιστον στα αγγλικά χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο. Στο σημείο K, στην παράγραφο μάλλον K, K, λέγεται οι προκλήσεις οι οποίες μυφίστανται. Μα ποιες προκλήσεις ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ ασαφής η διατύπωση εδώ πέρα. Πρέπει συγκεκριμένα να αφαιρθείτε σε κάποιες προκλήσεις. Πάντα θα υπάρχουν προκλήσεις αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο. Δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τι ακριβώς θέλετε να πείτε με αυτό το σημείο. Λάινεν. Ο Λάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον συνάδελφο Ράγκελ, διότι τις τελευταίες 800 ώρες έχουμε προσεγγίσει ένα τον άλλον, μπορεί και τις τελευταίες 18 ώρες μέχρι αύριο το πρωί δηλαδή, να τα καταφέρουμε ακόμα σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα ήταν ότι ο τίτλος της έκθεσης δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το περιεχόμενό της. Ο τίτλος ήταν «Εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας» όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η λέξη «εφαρμογή» σημαίνει ότι εξετάζει κανείς πόσο έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τα δικαιώματά μας, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Η έκθεση όμως έχει ξεπεράσει τα όρια αυτά, παρουσιάζει νέες ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συνθήκη σε κάποια μελλοντική συνταγματική συνέλευση. Ε, χαίρομαι που με τη συμβιβαστική πρόταση Β έχουμε βρει έναν συμβιβασμό το οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση του Προέδρου της Επιτροπής, ε, του Συμβουλίου και ε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ήμασταν κατά του να γράφουμε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να εκλέγεται άμεσα. Τώρα έχει αφαιρεθεί το σημείο αυτό και πριν ε, λέγαμε ότι η επόμενη συνταγματική συνέλευση θα πρέπει να επανεξετάσει, να σκεφτεί, αλλά βρήκαμε ότι και αυτή η διατύπωση ήταν υπερβολικά ισχυρή. Την κάναμε πιο ήπια. Κατόπιν έχουμε τη συμβαστική πρόταση F. Και συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο Σιουπφλίν ότι δεν θέλουμε δύο ειδών επιτρόπους με και χωρίς χαρτοφυλάκιο. Το θέμα είναι με τους αντιπροέδρους να έχουμε κάποιους ευρύτερους θεματικούς τομείς. Στην τροπολογία 57 το έχουμε διατυπώσει αυτό. όπου αναφερόμαστε στις αρμοδιότητες της Κομισιόν και και τις θεματικές ενότητες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Το θέμα είναι δηλαδή πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά των επιτρόπων. Κατόπιν έχουμε τη συμβαστική πρόταση ε ή πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. θα πρέπει να σκεφτούμε αυτήν ε, την πλειοψηφία των δύο τρίτων σε περίπτωση πρότασης μορφής προς την Κομισιόν. Θα πρέπει δηλαδή να είναι δυνατόν να μειωθεί αυτή η πλειοψηφία, αλλά το να αναφερόμαστε στην απόλυτη πλειοψηφία χωρίς να συζητήσουμε τις συνέπειες μας φαίνεται λάθος. Και τι εννοώ με αυτό. Είμαστε διαφορετικό κοινοβούλιο από τα εθνικά κοινοβούλια. Πολλοί το γνωρίζουν. Με απόλυτη πλειοψηφία και με το μάτι στα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών, δεν μου φαίνεται σωστό να μπορούμε να έχουμε πρόταση μορφής ε, κατά της Κομισιόν χωρίς να προβλέπουμε και τις συνέπειες. Εάν δηλαδή δεν έχουμε ε, κομισιόν θα έχουμε κρίση στην Ευρώπη. Στα εθνικά συντάγματα όταν ε, δεν υπάρχει κυβέρνηση για κάποιο χρονικό διάστημα προκυρήσονται εκ νέου εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό, να το συζητήσουμε εις, βά Κύριε Ράγγελ, λοιπόν, ε, έχω υποβάλει μια πρόταση η οποία μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές η συνταγματική συνέλευση θα πρέπει να συζητήσει την πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 234. Θα πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η πλειοψηφία. Διότι Κάποιοι αναφέρθηκαν σε αυτές τις προτάσεις μορφής και τι μορφή θα μπορούσαν να έχουν στην Ισπανία και τη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αφήσουμε λοιπόν ανοιχτό το θέμα της πλειοψηφίας. Το αν θα πρέπει να είναι πλειοψηφία των δύο τρίτων. Κατόπιν απομένει το σημείο όμικρον. Να αναφερθώ στη συμβαστική πρόταση νη. Συμφωνήσαμε Ο κύριος Ράνιελ έχει αντίγραφο που έχει λάβει από τον συνάδελφο Μπρόκ, οπότε μπορεί να παρακολουθεί αυτά που λέμε. Το έλαβε κάπως αργά, αλλά δεν πειράζει. Στο εν, λοιπόν, θα ήθελα να πω... ότι έχουμε τον ε, συμβιβασμό που μπορούμε να δεχτούμε. Το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει καταφέρει οι βουλευτές ε, κατά ε, την ε, υπογραφή συμφωνιών να μπορούν να είναι παρόντες και στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας θέλουμε και εμείς να το έχουμε αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε διατλαντική συμφωνία, εφόσον τα μέλη του Κογκρέσου μπορούν να συμμετέχουν από πλευρά της Αμερικής, τότε θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να συμμετέχουμε. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο πλαίσιο της αμοιβαιότητα. Τέλο, όσον αφορά το συμβασμό όμικρον. Δεν ξέρω ποιε είναι οι εμπειρίες ε, άλλων συναδέρφων όσον αφορά το πρόγραμμα που μας υποβάλλει η Κομισιόν, αλλά στην τροπολογία 103 Είπαμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξερευνά τη δυνατότητα να εκπονεί και να παρουσιάζει το δικό του πολιετές πρόγραμμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα σχέδιο της Κομισιόν και ένα σχέδιο της Κομισιόν. Έτσι, και ένα από το Κοινοβούλιο, συγγνώμη, και έτσι θα μπορεί να έχει περισσότερο βάρος η πρόταση, η θέση του Κοινοβουλίου. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε το πρόγραμμα της Κομισιόν, θα μπορούμε να εργαζόμαστε με βάση το δικό μας και όχι με βάση το δικό τους. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική πρόταση. Πάντως, κατά τα άλλα, έχουμε καταφέρει να βρούμε συμβασμού σε πολλά σημεία. Ευχαριστώ. Θα ε, σε ευχαριστούμε, κύριε Λάινεν. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρόκ. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες που σχετίζονται με δικές μου τροπολογίες, μπορώ να συμφωνήσω με τις προτάσεις του συναδέλφου Ράγγελ. Όσον αφορά την ε, τροπολογία F θα ήθελα να διαφωνήσω με τον συνάδελφο Λάινεν ε, ότι αν έχουμε θεματικές ενότητες θα πρέπει να υπάρχει και σχετική ιεράρχηση. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη διάρθρωση. Κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε στην κατάσταση όπου θα υπάρχουν λιγότεροι επίτροποι από ό,τι κράτη-μέλη. Και 28 επίτροποι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου, όχι όμως απαραίτητο και δικό τους χαρτοφυλάκιο. Μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν σε κάποια θεματική ενότητα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει λοιπόν η απαραίτητη διάρθρωση, διότι αλλιώς δεν θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Ε, είχαμε το Ιρλανδικό δημοψήφισμα όπου αναφερόταν η μείωση ε, του αριθμού των επιτρόπων. Εγώ πιστεύω ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπροσωπείται. Διότι έτσι δίδεται και η δυνατότητα στο πρόεδρο της Επιτροπής ε, να αναδιαρθρώσει την Επιτροπή εάν κάποιος επίτροπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μπορεί να ορίσει κάποιον άλλον. Είναι ένας τρόπος αυτός ο πρόεδρος της Επιτροπής να επιβάλλει κάποιες αρχές. Και Πιστεύω ότι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να βρει έναν κατάλληλο συμβιβασμό, διότι τελειώς θα αποτύχει. Αν έχει οι 28 επιτρόπους και κατακαιρματισμό των ε, χαρτοφυλακίων όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό στηρίζω αυτά που έχει καταγράψει εδώ ο συνάδελφος Ράγγελ. Συμφωνώ δηλαδή με την τροπολογία F. Και Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτή αν θέλουμε να υπάρχουν δυνατότητες διεύθυνσης. Και απαιτείται από τα κράτη-μέλη να προτείνουν ικανούς ανθρώπους για την Κομισιόν. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς επιτρόπους να έχουμε έτσι η βελτίωση της ποιότητας. Είμαι απόλυτος πεπισμένος για το θέμα αυτό. Άλλη μια παρατήρηση αφορά την συμβαστική τροπολογία N. Είμαι κλασικός υποστηριχτής του διαχωρισμού των εξουσιών. Δεν θα ήθελα να συμμετέχω στι διαπραγματεύσει ε, τη εκτελεστική ουσίας αν πρέπει τελικά να εγκρίνω το αποτέλεσμα. Διότι έτσι δεν υπάρχει σωστό έλεγχος. Θα ήθελα σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε να είμαι ελεύθερος να πω ναι ή όχι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν επί ένα εξάμεινο συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις είναι επιθυμία κάθε κοινοβουλίου να συμμετέχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά εγώ μπορώ μόνο να συμβουλέψω το αντίθετο. Όσοι καθοδηγούν τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις διαπραγματεύσεις, να τις καθοδηγούν, να λογοδοτούν και σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση διαπραγματεύσεις, ε, εκφράζει την ε, θέση του κατά την επικύρωση. Αυτά είναι τα κλασικά καθήκοντα ενός Κοινοβουλίου και γι' αυτό δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος με το συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ στο τελευταίο του σχόλιο. Συμφωνώ και με τον κύριο Αντζέλ ότι η πρόταση Γκερέρο το Κοινοβούλιο να συντάσει ετησίωση κάθε ορισμένα χρόνια το δικό του νομοθετικό πρόγραμμα είναι λανθασμένη. Πιστεύω ότι αν επιλέγαμε αυτή τη λύση ε, κάποια στιγμή θα χρειαζόταν να εγκαταλείψουμε διότι θα μας απασχολούσε πάρα πολύ χρόνο από τα άλλα μας καθήκοντα, ε, τα νομοθετικά μας καθήκοντα, τα καθήκοντα κοινοβουλευτικού ελέγχου κλπ. Χρειαζόμαστε ασφαλώς ένα κοινοβούλιο προσανατολισμένο στη στρατηγική για το μέλλον. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τη σύνταξη νομοθετικών προγραμμάτων. Θα μπορούσαμε να το πετύχουμε ε, με την επιλογή κατάλληλων ηγετών και με σοκαλής δουλειά σε επιτροπές. Σε ό,τι αφορά τα clusters, Νομίζω ότι υπάρχει μια φυσική ιεραρχία εντό τη Κομισιόν, το οποίο σημαίνει ότι στα κλάστα θα πρέπει να προεδρεύουν αντιπρόεδροι. Η διαδικασία είναι σαφής. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κομισιόν εμφανίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο ας πούμε και μας εκθέτει το πρόγραμμά του για το κολέγιο, για την ε, ε, ο, της Κομισιόν. και ζητώντας μας ε, να φέρουμε σε περαστής ε, ακροάσεις με βάση αυτό το πρόγραμμα. Και εκεί το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει την άποψή του για το κατά πόσον αυτό το πρόγραμμα, το πλάνο είναι καλό ή όχι. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Μπαρόζο να εξετάσει το ανεχόμενο της δημιουργίας clusters το 2009, αλλά αρνήθηκε. Όπως επίσης αρνήθηκε να ασκήσει το δικαίωμα του, το δικαίωμα που έχει για ανασχηματισμό της Κομισιόν κατά τη διάρκεια της θητείας. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Αν είχε ασκήσει αυτό το δικαίωμά του, αυτή την εξουσία του, θα την είχε εμπεδώσει. Και η Κομισιόν θα ήταν και πιο αποτελεσματική. Θα υποστηρίξω τη συμβαστική πρόταση F υπό την προπόθεση ότι θα στηριχθεί και η συμβαστική πρόταση G που ζητά να επανεξεταστεί στην επόμενη διάσκεψη το θέμα της, του μεγέθους της Κομισιόν. Γιατί δεν πιστεύω ότι τα καταφέραμε με τη σύνδεξη της Λισαβόνας. Είναι άχρηστο να προσπαθούμε να επιβάλλουμε στο Συμβούλιο να δεχτεί από μόνο του την κυκλική αναλλαγή των επιτρόπων. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας διάσκεψης. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετήσουμε την πρόταση της επικοδομητικής πρότασης μορφής. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα να απολύσει τον πρόεδρο της Κομισιόν υπό την προπόθεση ότι θα έχει βρει έναν αντικαταστάτη. Τώρα, αν αυτό θα πρέπει να γίνει εδώ ή στην διακυβερνητική διάσκεψη, αυτό δεν το ε, γνωρίζω, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν αυτούς, αυτές οι συμβαστικές προτάσεις, όπως έχουν. Και ο κύριος Σέφνερ, τελευταίος ομιλητής. Eh, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ. Α, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για όλες ε, τις προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών. Η δική μου πολιτική ομάδα βρίσκει καλές τις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συζήτηση δεν έχει γίνει ακόμα, αφορά τις συμβαστικές FG και H. Τι θα γίνει λοιπόν όσον αφορά το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ε, παρούσα πρόταση την αντιλαμβάνομαι ως εξής. Είχαμε την αρχική πρόταση με τους επιτρόπους άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παραμένει ως η μοναδική πρόταση, συνεχίζει όμως να αποτελεί μια δυνατότητα μαζί με άλλες δυνατότητες όπως είναι αυτή των θεματικών ενωτήτων εντός της Κομισιόν, των κλάστερ. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλύτερο, στο ιδανικό μέγεθος της Κομισιόν και στην καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών. Πιστεύω ότι είναι καλό να παρουσιάζουμε τις δυνατότητες χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα όμως να κάνω την εξή έκκληση. Στη συμβαστική πρόταση F να συμπεριλάβουμε την πρόταση σημαντικής μείωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που θα μας λείτωνε από τη λύση των Επιτρόπων χωρίς χαρτοφυλάκιο. Καταλαβαίνω ότι δεν σου αρέσει το μοντέλο αυτό. Υπάρχουν και λόγοι που κάθε χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να έχει έναν επίτροπο. Εγώ όμως δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο και έχω ανησυχίες, έχω επιφυλάξεις απέναντι και στην πρόταση με τα κλάστερ, με τις θεματικές ενότητες και στην πρόταση με τους επιτρόπους χωρίς χαρτοφυλάκιο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την πρόταση αυτή ως τρίτη δυνατότητα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας μια συνταγματική συνέλευση. Κάτι που ο Παύλο Ραγχέλ προβλέπει και για άλλες προτάσεις. Αυτή είναι η πιο σημαντική παρατήρηση. Θα ήθελα όσον αφορά την ψήφο μη εμπιστοσύνη στην πρόταση μορφή να συμφωνήσω με τον ε, Λάινεν. Είχαμε τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και καταλάβαμε ποιοι λόγοι αντίκυνται στην πρόταση αυτή. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε εδώ ως πρόταση, ως κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να συζητήσει η επόμενη συνταγματική συνέλευση. Και γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση του Γιώλαϊνεν, με την τροποποίηση που προτείνει. Κατά τα άλλα μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες. Σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνούμε μάλιστα πάρα πολύ. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις. Σας ακούσουμε τώρα την απάντηση του κυρίου Ρανζέλ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να απαντήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, δύο σημεία τα οποία έχει θίξει ο κύριος Σέπφλιν που μου προκαλούν κάποιες ανησυχίες. Νομίζω ότι η σημαστική και είναι σαφές ότι μιλάμε για την πρόκληση της διαφάνειας. Πρόκληση της διαφάνειας και αυτό μπορεί να επιληθεί με την έγκριση νέων κανόνων. Νομίζω ότι είναι σαφής η διατύπωση. Τώρα, ο όρο specificity, ιδιαιτερότητε, όντω μπορεί να είναι κάπω αόριστο, αλλά ποια είναι η βασική ιδέα εδώ πέρα. Με τη συμβαστική F, G και H έχετε μια ενότητα συμβαστικών προτάσεων. Και η βασική ιδέα πίσω από αυτέ είναι ότι όλα τα μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Όλε οι προσεγγίσεις ουσιαστικά. Ενδεχομένω λοιπόν να είναι κάπως περιττή η αναφορά που γίνεται εδώ πέρα. Στη συμβαστική F λέγεται με την επιφύλαξη να μπορείτε να, να διορίζετε μάλλον ένας επίτροπος ανακράτος μέλος. Αυτό όμως δεν αναφέρεται στη συμβαστική H και γι' αυτό το λόγο λέγεται ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών για να επιτυγχάνεται η ευκταία ισορροπία. Ουσιαστικά αυτό κρύβεται πίσω από τα όσα λέμε αυτή τη στιγμή, τα όσα λέγονται ουσιαστικά στην ε, συμβαστική πρόταση F, ότι κάθε χώρα θα έχει τον επίτροπό της. Αυτό θέλουμε ουσιαστικά να διασφαλίσουμε και στην ε, άλλη πρόταση, που απλώς λέμε όλα τα συμφέροντα των κρατών μελών, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι επίτροποι δεν εκφράζουν εθνικά συμφέροντα, λειτουργούν για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε όχι μόνο ουδετερότητα, αλλά και αντικειμενικότητα, προάσπιση δηλαδή όλων των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω πάντως ε, να υιοθετήσω εδώ πέρα μια διατύπωση πιο συγκεκριμένη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό τώρα για μένα είναι το εξή. Πρώτον, συμβαστική F και το πρόβλημα του χαρτοφυλακίου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να διατυπώσω τα πράγματα καλύτερα από τον κύριο Μπρόκ. Και ο κύριος Χέφνερ νομίζω ότι παρουσίασε τα πράγματα πολύ καλά. Η ιδέα εδώ πέρα δεν είναι να αναδιοργανώσουμε εντελώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες λύσεις για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι λύσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν πρώτον κλάστρες θεματικές ενότητες υπό έναν αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, η ιδέα του να έχουμε επιτρόπους με χαρτοφυλάκιο και άνευ χαρτοφυλακίου και δεχομένως τρίτον να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα μείωσης ή εκπεριτροπής εκπροσώπησης προβλέπεται η συνθήκη της Λισαβόνας. Και λέμε παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και την δυνατότητα αυτοδιοργάνωσης, αυτοργάνωσης μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ εμπνέουμε από τη γερμανική πραγματικότητα και να προβλέψουμε απλώς αυτή τη δυνατότητα. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχω πάρα πολλές ελπίδες να σας πείσω, πάντως το σύστημα επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου θα ήταν το καλύτερο δυνατό για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί κάθε κράτος μέλος θα έχει την επίτροπό του κατά αυτόν τον τρόπο. Οι επίτροποι άνευ χαρτοφυλακίου είναι απόλυτα ελεύθεροι να μελετήσουν πιο άντα και καλύτερα τα χαρτοφυλάκια των άλλων επιτρόπων και επίσης οι επίτροποι αυτοί μπορούν να έχουν αρμοδιότητες εκπροσώπησης παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς και επίτροποι με χαρτοφυλάκιο και επίσης θα μπορέσουμε με τους επιτρόπους άνευ χαρτοφυλακίου να έχουμε ένα σύστημα εκπεριτροπής. Πολύ φοβάμαι ότι με το σύστημα των κλάστερς τελικά θα έχουμε τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουν αντιπροέδρους επιτρόπους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τα κλάστερ θεματικές ενότητες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επίτροποι από τις υπόλοιπε χώρες θα βρεθούν με υποδέστερες αρμοδιότητες. Νομίζω ότι με το σύστημα επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου τα πάντα είναι απόλυτα διαφανή. Ξέρει ένα επίτροπο ότι τα πέντε πρώτα χρόνια μπορεί να μην έχει χαρτοφυλάκιο, αλλά θα, τα έχει, θα το έχει για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα χωρών διαφορετικά, οι μεγάλες χώρες, οι οποίες θα έχουν επιτρόπους αντιπροέδρους με τα σημαντικότερα θέματα οργανωμένα σε κλάστρες, θεματικές ενότητες, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες, οι μικρότερες δηλαδή χώρες, θα έχουν θέματα τα οποία δεν θα είναι τόσο σημαντικά. Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε νέον Πορτογάλο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι θα έχουμε πρόεδρο από το Λουξεμβούργο, λέει ο κύριος Ντάφα. Λοιπόν, διατρέχουμε πάντως τον κίνδυνο αυτό. Ξέρετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ήθελε να διοργανώσει ένα σύστημα εκπεριτροπής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες όλα τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτό επιτυχάνεται καλύτερα με το σύστημα των Επιτρόπων Άνευ Χαρτοφυλακίου. Όχι ενδεχομένως με την εκδοχή που πρότεινε ο κύριος Μπροκ, αλλά τουλάχιστον με τη δυνατότητα αυτού του ανασχηματισμού και κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και η αρμοδιότητα εξουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έπειτα κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι δεν συμφωνώ καθόλου με τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ανέκαθεν ήμουνα κατά μια τέτοια δυνατότητας. Ωστόσο, εισάκουσα ένα άλλο επιχείρημα. Το Αμερικανικό Κογκρέσο για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσει που έχουμε εμεί για ένα σύστημα ελεύθερων συναλλαγών, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ή μάλλον να έχουν οι Αμερικάνοι μέλη του Κογκρέσου τα οποία να συμμετέχουν στι διαπραγματεύσει αυτέ. Μπορούμε λοιπόν εμεί αυτό να το δεχτούμε στα πλαίσια τη αμοιβαιότητα. Δηλαδή, όταν οι διεθνεί μα εταίροι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται με μέλη του Κοινοβουλίου του, τότε θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε επίση όρει. Αν όμω δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο για του εταίρου μα, τότε να μην προβλέπετε ούτε για μα. Ναι, ναι. Αναφέρομαι για αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων, αυτό που μας είπε ο κύριος Μορέιρα, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, γιατί παρακολουθεί όλες τι σχετικές διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις διεθνείς δηλαδή συμφωνίες που συνάπτουμε με τρίτες χώρες. Πάντως, η αρχή, η ρήτρα της αμοιβαιότητος μας δίνει τη δυνατότητα να δεχθούμε το επιχείρημά σας αυτό. Καταλαβαίνω ότι προφανώς θα πρέπει να εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, να εκπροσωπούνται για παράδειγμα βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου. Εγώ πάντως ε, προτιμώ τη μέθοδο John Walks και να αφήσουμε περισσότερο τον έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω να είμαι κάπω ε, τη παλαιάς σχολή. Ένα άλλο σημείο τώρα. Το θέμα της πλειοψηφίας. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην απόλυτη πλειοψηφία και τα δύο τρίτα της μελλοντική Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 376 μέλη, αυτό είναι που πρότεινα. Απόλυτη πλειοψηφία λοιπόν των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όχι αυτών οι οποίοι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Δεν θα πούμε 62 ή 60% 58%. Και έχουμε και την ρήτρα αυτή που δεν είναι η επικοδομητική πρόταση μομφής, αλλά Έχουμε εδώ πέρα τη διατύπωση του κυρίου Ντάφα, διασφάλιση της σταθερότητας και της λειτουργίας του συστήματος. Νομίζω ότι είναι αρκετά λογικό αυτό το οποίο προτείνουμε και νομίζω ότι αυτό τον στόχο θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά την απόλυτη πλειοψηφία των μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι αυτών που είναι παρόντες και ψηφίζουν. Απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μολονότι πρόκειται για απόλυτη πλειοψηφία, ουσιαστικά είναι μια ειδική πλειοψηφία, ενισχυμένη πλειοψηφία, όταν μιλάμε για 376 μέλη. Θα προσπαθήσω να επεξεργαστώ τις προτάσεις σας και να βελτιώσω κάπως τη διατύπωση σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις, ωστόσο πιστεύω ότι η γενικότερη διευθέτηση που έχουμε πετύχει στην F, G και H θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και ότι η συμβαστική πρόταση I θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Μολονότι αν στην F, G και H υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης της διατύπωσης, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, θα επεξεργαστώ τα σημεία αυτά και σήμερα αργότερα ή αύριο το πρωί νωρίς θα μπορέσουμε πάλι να συνομιλήσουμε για να δούμε τελικά αν συμφωνούμε, αν έχουμε καταλήξει σε μια τελική συμφωνία. Σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κύριε Πρόεδρε, αλλά ξέρετε ότι ε, καθυστέρησα στη χώρα μου δύο ολόκληρες ώρες, η πτήση μου δηλαδή, γιατί είχαμε μια απίστευτη κακοκαιρία στην ε, Πορτογαλία. Απίστευτη λοιπόν κακοκαιρία η οποία καθυστέρησε κατά δύο ώρες την πτήση μου. Δεν είναι τόσο δραματικό αυτό, αλλά τουλάχιστον έφτασε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε που ε, ασχοληθήκατε με όλα αυτά τα ζητήματα και σχετικά σύντομα. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ερωτήσεις. Η κυρία Γκουρμάη θα πάρει το λόγο. Θα θυμάστε ότι σε έκτακτη συνεδρίασή μας είχαμε συζητήσει για το ζήτημα αυτό και είχαμε πει ότι το πεδίο εφαρμογής που αφορούσε μόνο την ώρα των ερωτήσεων θα πρέπει να διευρυνθεί και να αφορά γενικότερα τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τις γραπτές ερωτήσεις. Ακούσαμε και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεύκοβιτς και στη συνέχεια, μετά από μια επιστολή της 21ης Ιανουαρίου βάσει της Συμφωνίας Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβουλευτήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν τροποποίησης στον υποεξέταση κανονισμό. Τρεις τροπολογίες κατατέθησαν και 36 τροπολογίες από τους Νταφ Χέφνερ και από την κυρία Γκουρμάη. Έχετε το λόγο κύριε Γκουρμάη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι τηλεγραφική. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνεδρίασης ε, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων και πήρα και διάφορες απόψεις ε, από μέλη, θετικά, θετικά σχόλια γενικά. Να σας πω τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και να σε ενημερώσει και για κάποιες πρόσθετες αλλαγές. Σε ό,τι αφορά το χρόνο ερωτήσεων, ε, έχουμε δύο συμβαστικές τροπολογίες για να καλύψουμε τις προτάσεις του Άντριου Νταφ. Ευχαριστώ πολύ Άντριου. Αυτές οι δύο συμβαστικές προτάσεις έχουν στόχο να ξεκαθαρίζουν τη σχέση μεταξύ κανόνων και παραρτήματος. Ε, κυρίως ε, η αλλαγή αφορά τις πρόσθετες ερωτήσεις, συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ε, σύμφωνα με τον κύριο Νταφ, οι συμπληρωματικέ ερωτήσει θα μπορούσαν να γίνονται δεκτέ με, πιο με πιο αυτόματο τρόπο, υπό την προπόθεση ότι συνδέονται με την αρχική ερώτηση. Αυτό θα έκανε πιο ζωντανή τη συζήτηση, εξασφαλίζοντα ότι κανένα μέλο δεν θα, θα μπορούσε να καταχραστεί αυτή τη διάταξη, έτσι ώστε να κάνει ερώτηση για ένα διαφορετικό θέμα, δεύτερη ερώτηση για διαφορετικό θέμα. Υπάρχει όμω και ένα θέμα το οποίο δεν, δεν καλύπτεται από την τροπολογία ε, ο κ. Νταφ θέλει να αναφέρει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως ενδεχόμενο συμμετέχοντα στο χρόνο ερωτήσεων. Όμως ε, αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη, οπότε η πρόταση είναι αυτή η δυνατότητα να παραμείνει ανοιχτή για το μέλλον. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για αυτό το θέμα. Οπότε δεν διαφωνώ με αυτή την τροπολογία, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, έχοντας σκεφτεί το θέμα και μετά από συζητήσεις όμως με τις υπηρεσίες μας δεν θα χρησιμοποιούσα ε, τον εσωτερικό κανονισμό προκειμένου να προωθήσω ένα τέτοιο πολιτικό μέτρο. Ίσως θα έπρεπε αυτό το θέμα να ρυθμιστεί σε συνεργασία με τα άλλα όργανα. Το ίδιο και με τη συμπερίληψη του Συμβουλίου στο χρόνο ρωτήσεων διότι κάτι τέτοιο δεν προορίζεται από τι συνθήκε, ούτε έχει, έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε προτείνω να διαγράψουμε την αφορά στο Συμβούλιο ε, μέσω μιας προφορικής τροπολογίας και να μην συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα στον εσωτερικό κανονισμό. Παραμένω όμως ανοιχτή για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Τώρα, πρόταση Hefner. Είναι ενδιαφέρουσα, το είχα και εγώ σκεφτεί παλιότερα. Ε, προβλέπει την, το διαμοιρασμό του χρόνου, όμως ε, εγώ προτείνω να κρατήσουμε το σύστημα τελικά που έχουν προτείνει. Ε, έτσι ώστε όλα τα μέλη να είναι ισότιμα. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σαφές, ε, πιο ξεκάθαρο. Τέλος, να σας ενημερώσω ότι σκοπεύω να υποβάλω δύο προφορικές τροπολογίες τεχνικής περισσοτροφήσεως, σύμφωνα με τις οποίες οι τροποποιημένοι κανόνες θα μπουν σε εφαρμογή στην τη Δετάρτη την της πρώτης συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές και δεύτερον θα ε, επαναξιολογηθεί η δυνατότητα, μάλλον το σύστημα επιλογής των μελών ε, που υποβάλλουν ερωτήσεις ένα χρόνο μετά την ε, έναρξη εφαρμογής του. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ερωτήσεις, Έχουμε ένα όριο αναμήνα, τιμή υπέρ ενός μεικτού συστήματος, σύμφωνα με, το, με τη Βουλή των Κοινοτήτων, με το σύστημα της Βουλής των Κοινοτήτων. Οι ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Αν κάποιος θέλει να υποβάλει περισσότερες ερωτήσεις, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνει με προσωπική παρουσία στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Και αυτό θα αξιολογηθεί ένα χρόνο μετά από τη ε, διάσκεψη των Πρόεδρων. Μετά έχω και την τροπολογία 32 δική μου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Είναι σημαντικό να έχουμε feedback στην προετοιμασία, οπότε περιμένω και, το, ε, και τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκουρμά, ήσασταν πολύ σύντομη. Κυρία Λεγκρίπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γκουρμά, για την έκθεσή της, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, εξορροπημένη και που ουσιαστικά έχει ως στόχο να τροποποιήσει το άρθρο 116 και το παράθυμα 2 και τηρεί τις αποφάσεις ε, κατευθυντήρες γραμμές της διάσκεψης των Προεδρών, αλλά και τις παρατηρήσεις όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να συνάδει όλο και περισσότερο ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό ουσιαστικά συνάδει με την ιδέα της χρηστής διακυβέρνησης και αυτός ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο ρόλος της δικής μας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συμφωνώ με τα α και β, τροπολογίες α και β της κυρίας Γκουρμάη, που κατά την άποψή μου ε, όντω ανταποκρίνονται σε αυτά τα δύο κριτήρια, να συνάδει ο κανονισμό μα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και να ακολουθούμε κάποιε ορθέ πρακτικέ και να διερευνούμε μια καλύτερη διαχείριση των κοινοβουλευτικών εργασιών. Ωστόσο, όσον αφορά τι γραπτέ ερωτήσει, αυτές θα πρέπει να κατατίθενται το απαραίτητο το κατάλληλο μάλλον χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται στη Σύνοδο δηλαδή την ώρα των ερωτήσεων να κατατίθενται αυτές οι γραπτές ερωτήσεις. Κάποιες αφιβολίες τώρα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την τροπολογία 8 του κυρίου Ντάφα που έχει ως ε, στόχο να συμπεριλάβει την δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ώρας των ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καταλαβαίνω την πολιτική, την πολιτική πτυχή που βρίσκεται πίσω από μια τέτοια πρόταση, πίσω από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ συμμετέχω σε μια αντιπροσωπεία στα πλαίσια της πολιτικής μου ομάδας που συνεχώς ζητούσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να έρχεται όσο δυνατόν πιο συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετέχει στις συζητήσεις και να μας ενημερώνει, αν μη τι άλλο, για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ισχυθούν οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό προφανώς όλοι το επιθυμούμε, ωστόσο γνωρίζουμε ότι η συνθήκη για λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεώνει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρήσεται και να δίνει εξηγήσει κατά τη διάρκεια της ώρας των προφορικών ερωτήσεων. Και επίσης, για να είμαστε πιο ακριβείς από νομικής πλευράς, δεν υποχρεώνεται να παίρνει το λόγο εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπώντας πιο συγκεκριμένα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν η τροπολογία 8 ως έχει αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες και μολονότι η πολιτική διάσταση της τροπολογίας αυτής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ωστόσο δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω με την τροπολογία αυτή ως έχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με την υφιστάμενη διατύπωση προτείνει ο κύριος Ντάφα. Αλλά υποστηρίζω τις δύο προφορικές τροπολογίες που μας πρότεινε η συγκήτριά μας και συμφωνώ και με το ευαίσθητο αυτό ζήτημα το οποίο θίξατε, ευαίσθητο για όλους μας. Ο αριθμός των ερωτήσεων που μπορούμε να υποβάλουμε ένα μήνα. Νομίζω ότι ο αριθμός βλέπετε εδώ πέρα είναι λογικός και δεν νομίζω ότι βάλει κατά του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης, αν θέλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριο Ντάφη, το λόγο. Ε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ την Ζήτα Γκουρμάη για την ε, επικοδομητική της ε, προσέγγιση και το πνεύμα συμβασμού που έδειξε. Θα στηρίξουμε τις ε, δύο συμβαστικές προτάσεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο ε, σημερινός Πρόεδρος λέει πολύ σωστά ότι δεν λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σωστό αυτό, διότι δεν τον έχουμε διορίσει εμείς, ούτε και μπορούμε να τον απολύσουμε. και λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσει σε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή μόνο. Ε, εγώ δεν έχω βρει καμία που θα μπορούσα να του θέσω για την προσωπική του ζωή. Αλλά παρόλο το γεγονό ότι επισήμω και τυπικά δεν λογοδοτεί σε εμά, έχει καθήκον να συνεργάζεται ειλικρινά μαζί μας. Επίσης, και θα το δούμε αυτό τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ε, όταν θα γίνει ε, ο, ο άνθρωπος που θα ε, ηγηθεί της Κομισιόν ότι, θα δούμε λέω, ότι η εξουσία του αυξάνεται. Συμβούλιο έχει την τάση να ε, επεκτείνει τις εξουσίες του. Και πολύ συχνά οι ηγέτες ε, ε, τεντώνουν την προσπαθούν να τεντώσουν τη συνθήκη της Λισαβόνας έτσι ώστε να τη φέρουν στα μέτρα τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να, μπορούν να, να μπορούμε να τους ζητούμε να εμφανιστούν ε, εδώ στο ε, κοινοβούλιο και να τους ε, περωτήσουμε. Τώρα, το κατά πόσον η, ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να ε, υπερβαίνει την de πραγματικότητα. Αν δεν την υπερέβαινε, δεν θα είχαμε καν οργανώσει τις ακροάσεις των επιτρόπων, των υποψηφίων επιτρόπων. Γιατί αυτές τις είχαμε συμπεριλάβει σε μια ε, συμφωνία πλαίσιο, τις συμπεριλάβαμε τελικά σε μια συμφωνία πλαίσιο. Είχαμε ξεκινήσει όμως ε, από μια κατάσταση την οποία δεν προβλεπόντουσαν από την νομοθεσία, από τη συνθήκη. είναι ένας τρόπος να σπρώξουμε τα πράγματα. Τώρα για τον αριθμό των ερωτημάτων έχω προτείνει την τροπολογία 15 ε, η οποία προβλέπει 6 ε, γραπτά ερωτήματα τον μήνα σε συνήθη θέματα συν μια ερώτηση προτεραιότητας. Ε, η συγγήτρια προτείνει την απάλληψη της διαφοράς μεταξύ ερωτημάτων προτεραιότητας και μη προτεραιότητας. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα. Νομίζω ότι η, ερώτηση η διάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι χρήσιμη. Πρέπει σίγουρα πάντως η οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή που θα κάνουμε να ε, αναθεωρηθεί ή να επανεξεταστεί μετά από ένα χρόνο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λίγα λεπτά έχουμε για την απάντηση κυρία Γκουρμά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας είχα δει, σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Έφνερ, έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Θα είμαι πολύ σύντομος, καθότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και εγώ ευχαριστώ στο όνομα της πολιτικής μου ομάδας για την έκθεση αυτή που πιστεύω ότι αποτελεί βελτίωση. Και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες ε, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Από την πλευρά της δικής μου πολιτικής ομάδας ε, θα ήθελα να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις. Καταρχάς ότι δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αυτό το σύστημα με τις κάλπες είναι το ιδανικό σύστημα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή ο χρόνος εν μέρη να μοιράζεται ανάλογα με τι πολιτικέ ομάδες. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι θα θεωρούσαμε βελτίωση να επιλέγεται ένα θέμα μήνα για την ώρα αυτή των ερωτήσεων. Δεν πιστεύουμε όμως ότι πρέπει απαραίτητα να έχουμε μόνο έναν θεματικό κύκλο. Εάν υπάρχουν διάφορα θέματα, μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε και να ε, έχουμε κάποιο χρόνο για τον ένα κύκλο και ένα κάποιο χρόνο για τον άλλον. Κατά τα άλλα, ο περιορισμός σε πέντε ερωτήσεις ε, πιστεύουμε ότι αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την παρουσία διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη είπα ότι το προβλέπω αυτό, δεν θέλω να τα επαναλάβω, διότι μας τελειώνει ο χρόνος και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις των άλλων συναδέρφων, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε καινοτομία να αποτελεί βελτίωση. επιδιώκουμε την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για την καθοδήγησή τη. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους, διότι όταν είναι κανείς εισηγητή, χαίρεται κανείς που ακούει τις διάφορες απόψεις, αλλά πρέπει να συγκεντρώσει ο εισηγητής τελικά τις απόψεις αυτές. Δώστε μου λοιπόν λίγο χρόνο. Πάντως ε, χαίρομαι που συμφωνείτε με τις προφορικές τροπολογίες μου. Δεν έκουσα καμιά αντίρρηση. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα καλό καινοτόμο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Είναι σημαντικό προνόμιο να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε αύριο το πρωί λοιπόν. Όπως σας είπα από τις 9 ως 9.30 θα έχουμε τη συνεδρία των στονιστών και κλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια από τις 9.30 ως 10.30 θα δούμε την τροποποίηση του άρθρου 90 του κανονισμού για τι διεθνεί συμφωνίες, καθώς επίσης και την τροποποίηση της Οργανική συμφωνίας σχετικά με το Μητρό διαφάνεια. και στη συνέχεια θα έχουμε την ψηφοφορία από τις 10.30 ω τις 11.30. Και στη συνέχεια θα καλύψουμε τα υπόλοιπα σημεία τα οποία προβλέπονται στην ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία, λύεται η συνεδρίαση. Αύριο το πρωί ξεκινάμε σε 9 με τους συντονιστές και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν στις 9.30 δύο αυτές εκθέσεις και στις 3.30 ψηφοφορίες.